On est prêt On est prête Oui, vous êtes très bien accompagné. Mesdames, Messieurs, je vous invite à gagner. Κυρίες αλλά και κύριοι, σας καλώ να καθίσετε στις θέσεις σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία σας. Με μεγάλη χαρά σας ε, υποδέχομαι στην τόσο σημαντική αυτή ακρόαση που οργανώνει η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε σχέση με το ρόλο των χρηματοπιστωτικών φορέων και την αρρωγή τους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, έχω δίπλα μου την κυρία Έιντερ Γουαρδία Σαβάλ και την κυρία Λία Νιριάντα που έχουν προετοιμάσει αυτή την ακρόαση, την ανταλλαγή αυτή απόψεων που θα περιλαμβάνει και συζήτηση και θα τους δώσω όσον ούπο τον λόγο. Έιντερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. <clears throat> Πάρα πολύ σύντομα γιατί όπως ε, έχετε διαπιστώσει η ημερησία διάταξη αυτής της ακρόασης είναι πάρα πολύ γεμάτη. Ήδη καθυστερούμε, επομένω θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σφιχτοί με τον χρόνο. Είναι φανερό ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών έχει συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν Πώ ε, μπορούμε να βελτιώσουμε τον αντίκτυπο του προπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον περίγυρό μα πώ μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τα σχέδια που αναπτύσσουν μικρομεσαίες επιχειρήσει στην περιοχή μα Και όταν μιλούσαμε για την οργάνωση αυτή τη ακρόαση για του χρηματοπιστωτικού πόρου και τη χρηματοδότηση μαζί με την ε, Λία, είχαμε αποφασίσει ότι θα πρέπει να εστιάσουμε ακριβώς σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και ιδίω να μεταφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές τράπεζες προώθησης οικονομίας μπορούν να χρηματοδοτήσουν σχέδια που εμπλέκουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι λοιπόν ο σημερινός στόχος και η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση για μένα να δω ότι είχαμε μια ημερησία διάταξη πιο ανοιχτή με πολλή συζήτηση που προβλεπόταν αλλά όσο οργανώναμε την ε, εκδήλωση αυτή ήταν όλο και περισσότεροι που θέλανε να συμβάλλουν και να συμμετάσχουν. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον για το έργο της Επιτροπής Προϋπολογισμού και γι' αυτό χαιρόμαστε πάρα πολύ για όλους τους ομιλητές που ήταν εδώ και θα δώσω το λόγο στην συναδελφό μου τη Λία. Παρακαλώ. Δεν πρόκειται να σας καθυστερήσω. Εδώ είμαι για να σας ακούσω περισσότερο. Νομίζω ότι είναι μεγάλη μας ευκαιρία να μπορούμε να κάνουμε αυτή την συζήτηση γιατί οι ΜΜΕ τόσο σημαντικές στην τοπική οικονομία και στην Ιρλανδία έχουμε ε, το 70% της εισφοράς αυτών στην οικονομία, την τοπική οικονομία. Όμως είδαμε ότι η απόρριψη της συνδανείων είναι τρομερή και αυτό της πνίγει της ΜΜΕ και για αυτό και περιμένω όπως και πώς να ακούσω σήμερα οπότε ευθύς αμέσως όπως ε, είπατε να συνεχίσουμε. Άρα δεν θυμάμαι το όνομά σα, δικό το Καλά, κύριε Ρούμπια, αν προσπαθήσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, ούτω ώστε να έχουμε αρκετό χρόνο για έρωτα απαντήσει. Πάμε τώρα λοιπόν στον τον πρώτο μιλητή. Πού να τον προφέρουν, τον Γουαρόν. Ε, είναι σε μια υψηλή θέση που εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την πρόσκληση και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα χρηματοδοτικά και χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία πρέπει να παρουσιάσουμε είναι κάτι το πρόσφατο. Είναι το πρώτο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που έχουμε αυτό το πλέγμα κανόνων για τα χρηματοοικονομικά τα οποία στο 8ο κεφάλαιο του κανονισμού καλύπτονται. Άρα προχωράμε μαθαίνοντας και έχουμε τις διάφορες αιτήσεις εκθέσεις και έχουμε και την μεσοπρόθεσμη ε, αναθεώρηση του πολιτούς πλαισίου, οπότε και έτσι θα κάνουμε έναν απολογισμό για τα πρώτα χρόνια της εμπειρίας αυτής της υπόθεσης. Ε, επομένως είπαμε ότι προχωρώντας μαθαίνουμε και έχουμε αυτόν τον ε, κανονισμό και όσον αφορά την κοινή διαχείριση έχουμε κάποιους κανόνες αλλά έχουμε πετύχει σύγκληση μεταξύ των ε, κανόνων που αφορούν την, και, την κεντρική διαχείριση αλλά και την συνδιαχείριση. Βέβαια πάντα επιδέχεται η σύγκληση ε, βελτίωση. Οπότε οι αρχές για αυτό ε, το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι κάποιες ενισχύσεις. Ενισχύσεις με τις οποίες δημιουργούμε την αγορά. Οπότε έτσι έχουμε τους κανόνες. Αλλά με τα χρηματοδοτικά και χρηματοοικονομικά ε, μέσα πάμε σε έναν τομέα ο οποίος ήταν ήδη ρυθμισμένος και υπάρχουν ήδη επομένω κάποιες πρακτικές στην αγορά όπως και κανόνες. Γι' αυτό και χρειάζεται ευελιξία. Οπότε αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι κάτι σαν σύμβαση μεταξύ της Επιτροπής που έχει την αρμοδιότητα την εφαρμοστική και τα άλλα θεσμικά όργανα, Συμβουλή Κοινοβούλια. Μας δίνετε την ευελιξία, αλλά θέλετε ε, να σας αναφέρουμε σχετικώς σε δακτά διαστήματα και να είμαι θα έχει υπόλογη σε σας. Και οπότε επί τη βάση αυτών των συνδικών της αγοράς θα πρέπει να δούμε, όταν γίνεται πρώτος για ένα νέο πολιτές πλαίσιο, να δούμε το ότι δεν είναι με τίποτα δυνατόν να κάνουμε προγνωστικά για την μέλουσα χρηματοδοτική, χρηματοοικονομική συγκυρία. Άρα, εσείς θέλετε να σας δίνουμε αναφορά, να σας ενημερώνουμε και επίσης Εάν κάποιο χρηματοδοτικό όργανο δεν αποδίδει, να το κόβουμε. Οπότε ευελιξία και απόδοση λογαριασμών και λογοδοσία. Πώς θα το καταφέρουμε, πώς θα έχουμε την ευελιξία. Έχουμε ένα πλέγμα βασικών κανόνων στον χρηματοδοτικό κανονισμό, στα άρθρα 139 και 140 προβλέπεται. Βασικοί κανόνες αυτοί όσον αφορά το να καλύψουμε ε, κάποιο κενό στην αγορά, να καλύψουμε επίσης κάποια προγράμματα ή έργα που είναι οικονομικά βιώσιμα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, προσθετικότητα, το πώς δηλαδή θα έχουμε, πώς θα λυκίσουμε ιδιωτικές επενδύσεις, να μην στρεβλώσουμε τον ανταγωνισμό, να έχουμε το αποτέλεσμα της βασικό επιχείρημα για να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα, αυτά τα εργαλεία, γιατί ε, θα πρέπει να υπάρχουν ε, αποτελέσματα που να κρατήσουν πάρα χρόνια Επίσης, το να μην ε, υπάρχει μετακύληση της ευθύνη και μία πίστοση του λογαριασμού να αρκεί. Ναι, εδώ μπαίνει ο, ο ρόλος του ΕΦΣΙ, του Ταμείου Σωτικών Επενδύσεων. Έχουμε πάρει 16 δις από την Τράπεζα Επενδύσεων. Αλλά εμείς είπαμε ότι ε, καλύπτουμε με τις εγγύσεις το 50% αυτής της πρικοδότησης, αυτής της ε, πίστοσης. Οπότε έχουμε αυτούς τους βασικούς κανόνες και σε κάτι επομένω πράξη έχουμε μία βασική έγκριση. Η βασική πράξη δεν φτάνει να καλύψει όλες τις λεπτομέρειες και τις παραμέτρους ε, από την αρχή. Οπότε εδώ πέρα μπαίνει ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο ρόλος της ευελιξίας. Άρα, πώς θα εξασφαλίσουμε αυτή την υποχρέωση λογοδοσίας. Έχουμε κάποιους δείκτες απόδοσης μεταξύ των οποίων είναι και η μόχλευση. Αυτό υπολογίζεται σχετικά εύκολα. Επίσης, έχουμε την δοκιμή της αγοράς. Υπάρχει ζήτηση πλευρά αγοράς για το χρηματοδοτικό εργαλείο που Ξεκινάμε. Ο, για όλα αυτά υποβάλλουμε εκθέσεις, αναφέρουμε σχετικά και υπάρχουν αξιολογήσεις κλπ. Όμως υπάρχει μια ετησία έκθεση όπου έχουμε ένα ολόκληρο κατάλογο από τις παραμέτρους του άρθρου 140 8 του κανονισμού. Όλα αυτά οφείλουμε να τα αναφέρουμε. Οπότε έχουμε και την αίρεσιμότητα όσον αφορά την συνέχεια της επίδοσης απόδοσης. Οπότε το πρώτο τεστ είναι όταν έχουμε την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, όταν ε, βλέπουμε, όταν τελειώνει το πρώτο μισό της ε, ζωής αυτού του οργάνου και θα πρέπει να δούμε ε, τι καλύπτει τις προσδοκίες μας και τι υπολείπεται από τα χρηματοδοτικά όργανα ή μέσα μάλλον. Οπότε θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν κάποια μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Και είπαμε ότι αυτά τα μέσα ή όργανα μπορεί να τα επιστρατεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άμεσα ή έμεσα από, να γίνει από κάποιους φορείς. Και εσείς ως νομοθέτες τα έχετε αυτά αναφέρει στον κανονισμό και ξεκινάτε με την ΕΤΕ και το Ίδρυμα Επενδύσεων τράπεζες και λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα κρατικά. Και θα δούμε κατά τη διάρκεια της ε, σημερινής ακρόασης ότι είτε το Ταμείο είτε οι Τράπεζα Επενδύσεων έχουν συγκριτικά πλειονεκτήματα. Η ΕΤΕ και το Ταμείο Επενδύσεων μπορούν να καλύψουν τα 28 κρατημέλη και να εξασφαλίσουν την μεγίστη γεωγραφική κάλυψη. Και αυτές οι εθνικές τράπεζες πρόθεσης ξέρουν τι ισχύει επιτοπίως. Είναι εταίροι των ε, αρχών διαχείρισης και ένα από τα προβλήματα που ακόμη έχουμε σε αυτή τη διαδικασία όπου μαθαίνουμε είναι το πώς θα γίνει ο κατάλληλος συνδυασμός αυτών των θεσμών για να αποδώσουν. Μιλήσαμε για τα ΜΜΕ προηγουμένως, οπότε έχουμε α, ε, αυτούς τους φορείς τους οποίους, τους οποίους εξουσιοδοτούμε να χρησιμοποιήσουν το χρηματοδοτικό μέσο και οπότε για τις ΜΜΕ ή θα πρέπει με, με εταιρικό κεφάλαιο να κινηθούν ή θα να πάρουν κάποια δάνεια αλλά ο επιλέξιμος, ο δικαιούχος μάλλον δεν είναι άμεσα η, η ΜΜΕ. Έχουμε κάποιους ενδιάμεσους ε, συνέδους, είναι εμπορικές τράπεζες. Για τη μικροχρηματοδότηση βέβαια έχουμε και άλλα ιδρύματα που δεν είναι τράπεζες, αλλά για τις ΜΜΕ υπάρχει το πρόβλημα των γραφειοκρατικών κοινοτικών κανόνων, γιατί έμεσα στη ΜΜΕ από μια, συνήθις, από μια συνήθη πρακτική που διέπουν την αγορά κλπ. Τώρα, θα πρέπει να δούμε το πόσο στεγανό είναι αυτό το πλαίσιο κανόνων και ποια είναι τα προβλήματα. Μέχρι τώρα, παρά το ότι είναι φρέσκο ακόμα αυτό το χρηματοδοτικό μέσο, ε, το ότι θα πρέπει να εξισορροπήσουμε από μία μεριά την, το συμβατό με την αγορά και από την άλλη μεριά την υποχρέωση λογοδεσίας. Να πούμε ότι στα περίπου καλά τα έχουμε πάει. Νομίζω ότι πετύχαμε ακριβώς γιατί προηγήθηκαν οι συμβουλές το ταμείο Επενδύσεων και της Τράπεζας Επενδύσεων. Αλλά επίσης και η στενή επαφή που είχαμε με τις Εθνικές Τράπεζες Πρώτης Οικονομίας. Ξέραμε επομένως πώς θα καταφέρουν τη σωστή ισορροπία. Δεν ξέρω αν θα σας ε, ε, εκπλήξει η συζήτηση ότι εδώ πέρα γίνεται κουβέντα για την διαφάνεια. Πριν φτιαχτεί το ρυθμιστικό πλαίσιο ξεκίνησε αυτή η προβληματική. Δεν είχαμε κανόνε. τώρα έχουμε να πλέγουμε κανόνων. Οπότε παρέχονται τις σχετικές πληροφορίες, ενημέρωση. Το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι, όπως είπαμε πριν, το ότι στηριζόμαστε σε τράπεζες και λοιπά ιδρύματα κρατικά. Είναι δηλαδή οι εταίροι μα επαγγελματίες. Ξέρουν τις πρακτικές της αγοράς ξέρουν τι αναγνωρίζει ο ιδιωτικός τομέας, τι θεωρείται σαν θεμητό, σαν νόμιμος παίκτη ε, σε αυτή την κατάσταση. Και έτσι και προχωράμε με αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Μιλάμε πάντα, δεν μιλάω για την οικονομία και τα οικονομικά προβλήματα, μιλάω για το ρυθμιστικό πλαίσιο. Και βέβαια θα πρέπει να παραδεχτώ και το που υστερούμε. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας το υπήν από πλευράς χρηματοοικονομικής και εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα πράγματα εδώ δεν είναι σαν τις ε, ενισχύσεις, είναι πιο περίπλοκα. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τις αρχές διαχείρισης. Για ένας από τους φραγμούς που υπάρχουν για να αξιοποιηθούν αυτά τα εργαλεία είναι το ότι κατά κυριαρχεί η φιλοσοφία, η κουλτούρα της ενίσχυσης, της επιδότησης. Ε, αυτό θα το καταφέρουμε, αλλά θέλει χρόνο να το αλλάξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά. Οπότε και εδώ, από πλευράς ελέγχου, δηλαδή Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, πάλι θα πρέπει να μάθουν οι ελεγκτικές αρχές. Να που μπαίνει η διαφάνεια. Έχουμε τις πληροφορίες, όπως είπατε στον κανονισμό, όπου θεσπίσατε τις σχετικές παραμέτρους που να συλλέξουν. Οπότε απόκειται σε εμά να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία και τις πληροφορίες. Δεν αρκεί η μόχλευση για να ζυγίσουμε τις επιδόσεις ενός εργαλείου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει το εργαλείο αυτό με την αγορά. Όμως η αξιολόγηση χρειάζεται και μια εμπειρογνωμοσύνη που σιγά σιγά όλοι μας την αποκτούμε. Άλλο πρόβλημα. Και όταν εμείς νομοθετούμε και όταν εσείς ε, κρίνετε θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, θα πρέπει να αυξήσουμε τη δυνατότητά μας να είμαστε όσο γίνεται πιο ακριβείς στο να επισημάνουμε ποιο πρόβλημα στην αγορά θέλουμε να καλύψουμε. Γιατί έχουμε κάποιους κλάδους ή τομεί που όντω χωλαίνει εκεί η τομει που όντω Υπάρχει πρόβλημα. Και δεν υπάρχει συνταγή επιστημονική γι' αυτό. Χρειάζεται αξιολόγηση. Χρειάζεται κανείς να λάβει υπόψη πολλές μεταβλητές. Αλλά το να κάτσει κανείς και να βρει ακριβώ το που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις να δει κανείς ποιο είναι το πρόβλημα, να το μετρήσει ακριβώς, να κάτσει και να δει ποιο είναι το κενό της χρηματοδότησης ε, για τις ΜΜΕ. Αυτό είναι δύσκολο. Από πού είναι. Από την πλευρά της προσφοράς, από τις τράπεζες είναι το πρόβλημα. Ή για το ότι δεν ε, υπάρχει υγιής, ε, αξιόπιστη, αξιόχρεη ζήτηση. Άρα να τη χρειάζεται να ξέρει κανείς καλά για να σχεδιάσει καλά το χρηματοδοτικό εργαλείο. Τέλος δε, θα πρέπει να διευρύνουμε τους διάβλους της χρηματοδότησης, της παροχής ας πούμε, όχι να φτιάξουμε καινούριου διάβλους, θα πρέπει να υπάρχει συνέργεια μεταξύ των υπαρχών των διάβλων, να δούμε αν θέλουμε να στηρίξουμε τις ΜΜΕ, γιατί έχουμε κάποια κέντρο κατευθυνόμενα προγράμματα και χρηματοδοτήσεις από εδώ, οπότε ακόμα και αν υπάρχει σύγκληση στα προγράμματα υπάρχουν ε, διαφορετικά σημεία που κανείς θα πρέπει να καλύψει. Υπάρχει συνδιαχείριση με τα διευθυντικά ταμεία, υπάρχει η πρωτοβουλία για τα ΜΜΕ που έχουν τους δικούς τους κανόνες και τώρα υπάρχει και το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, το ΕΕΦΣΙ. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συνδυάσουμε. Άρα είναι τα πράγματα περίπλοκα. Και αυτό αποδεικνύει ότι χρειάζεται πολύ και η τεχνική αρρωγή στις ε, αρχές της διαχείρισης σε αυτούς που τρέχουν τα έργα και τα προγράμματα. Τεχνική αρρωγή για αυτά τα προγράμματα κύριε. Ό,τι ρωτήσετε θέλετε μπορείτε να υποβάλλετε. Bien, merci, monsieur. Καλώς. Κύριε Διευθυντά, σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, έχουμε τώρα 10 λεπτά στη διάθεσή μας για ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων. Ο κύριος Φερνάντης. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την διοργάνωση αυτού του σεμιναρίου και θα ήθελα επίσης να ε, ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για αυτή την παρέμβαση. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Ήδη βρίσκονται σε φάση εκτέλεσης όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα. Για παράδειγμα, ε, ε, το Creative Europe, το χρηματοοικονομικό μέσα, μέσο ή το LIFE, το πρόγραμμα LIFE. Οπότε ρωτάω, σε σχέση με αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα, ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ. Και δεύτερο ερώτημα, γιατί υπήρξαν καθυστερήσει σε ό,τι αφορά τη θέση σε ισχύ αυτών των χρηματοδοτικών μέσων από την ε, πλευρά των κρατών μελών ε, διασφαλίζεται η ε, κατάλληλη απορρόφηση αυτών των μέσων, ώστε να μην υπάρχει άνισο κατανομή και άνιση διανομή αυτών των κονδυλίων σε ό,τι αφορά τις περιοχές. Και επίσης, έχετε προβλέψει ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της μόχλευσης και αυτή η μόχλευση όπως τώρα ε, διαγράφεται βρίσκεται εντός των ε, δικών σας προβλέψεων όπως είχατε κάνει. Ναι, πρέπει να θέλετε κάποιος σας να θέσει ένα ερώτημα. Ποιος θέλει να ξεκινήσει από εσάς. Ηλία, ναι, ευχαριστώ πολύ για την συμβολή σας. Για μένα είναι περισσότερο πως μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι είναι πιο προσβάσιμη αυτή η πληροφορία. Έχω την εμπειρία της δικής μου χώρας, αλλά ξέρω ότι είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα. Δεν έχουμε μια εθνική ε, τράπεζα αναπτυξιακού χαρακτήρα στην Ιρλανδία, που κάνει πολύ δύσκολο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε κονδύλια Πώς θα περάσουμε λοιπόν αυτό το σκόπελο, πώς θα ξεπεράσουμε αυτό το χάσμα. Υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αναφέρατε. Υπάρχουν ε, δυσκολίες ε, και τέλματα στα οποία καταλήγουν τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και η μικρομεσαία επιχείρηση δεν ξέρει περί πρόκειται. Επομένω, οι διαχειριστικέ αρχέ χρειάζονται να έχουν πια κάποια βοήθεια ώστε να παίρνουν την κατάλληλη πληροφορία για να δώσουν σε αυτού του ανθρώπου και να δημοσιοποιήσουν όλε αυτέ τις δυνατότητε γιατί δεν είναι γνωστέ. Η Έιτερ. Ναι, ευχαριστώ και εγώ πολύ. Σε, αυτό το πρώτο, σε αυτή την πρώτη παρουσίαση είδαμε ότι υπάρχουν ε, πολλές, ε, πολλά παρόμοια στοιχεία όπως και για τη συζήτηση που κάναμε για το ΕΦΣΙ, το σχέδιο Juncker. Πώς μπορούμε να δώσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες στις διάφορες αρχές, ιδίως τις περιφερειακές αρχές, ώστε να φτάσουμε αυτά στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ένας από τους φόβους που είχαμε ήταν ότι ακριβώς δεν υπήρχε η συσσωρευμένη πείρα με τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο κύριος Κερό είπε ότι η Κομισιόν προσπαθεί μαζί με την διαδικασία αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου, του πολιετούς πλαισίου, εργάζεται και για την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα είναι κάτι στο οποίο μπορείτε να απαντήσετε, αλλά ακριβώς προ ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η Κομισιόν για να μπορέσει να εξαλείψει τα προβλήματα τα οποία μπορούν να ανακύψουν τώρα με τη διαχείριση των χρηματοδοτικών εργαλείων και αν μπορείτε να πείτε σε περισσότερε λεπτομέρειε ποια είναι τα στοιχεία αυτά τα οποία δεν λειτουργούν αρκετά καλά, πού είναι τα προβλήματα που έχετε εντοπίσει και πώ προσπαθείτε να δράσετε ώστε αυτά τα εργαλεία να είναι πιο επωφελή στη δράση του. Χωρίς μικρόφωνο. Και εγώ θέλω να θέσω ένα του χωρι μικροφωνο και εγω θελω Έχετε την εντύπωση ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο που υπάρχει είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να επιτρέψει ταχείες ενέργειες και ταχείες και αποτελεσματικές επεμβάσεις στα θέματα αυτά. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή με τις τωρινές συγκυρίες έχει ένα τεράστιο πλωστάσιο κανόνων και ρυθμίσεων που δεν είναι πάντα απόλυτα συμβατές και μεταξύ τους. Έχετε λοιπόν την εντύπωση κύριε Κερομουσό ότι τα εργαλεία αυτά είναι εργαλεία τα οποία είναι καλώς θεσπισμένα, είναι κατάλληλα για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Και αν δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα, ξαναδώσω στον ομιλητή του κύριο Κερομισό το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν μπορώ να ξεκινήσω με την τελευταία σας ερώτηση. Όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε επαρκώς στο ρυθμιστικό πλαίσιο στοιχεία ευελιξίας. Δηλαδή, αν έχουμε ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, αρκεί το πρόγραμμα μας να προβλέπει να έχει αυτή τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο και πολλές φορές τα θέματα υποδομών, καινοτομία, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενεργειακής απόδοσης προβλέπεται η δυνατότητα να γίνουν τέτοια εργαλεία. <clears throat> Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τη νομική βάση για να μπορέσουμε να προβούμε στη δημιουργία ενός τέτοιου εργαλείου. Έχουμε καταρχήν βάσει τον κανόνα μας μία εκ των προτέρων εξάντε ανάλυση. Σε περιπτώσεις έκτατης ανάγκης μπορούμε να απλοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά πάντα πρέπει να προβούμε σε μία ανάλυση η οποία θα μας επιτρέψει να καταλάβουμε τι είδους παρέμβαση πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Έλεγα προηγουμένως στα συμπεράσματά μου ότι γενικά έχουμε πετύχει μια καλή ισορροπία. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα και να κάνουμε το λεγόμενο fine tuning, να εξευγενήσουμε λιγάκι τις ρυθμίσεις μας και να καταλύσουμε τα στεγανά που υπάρχουν ανάμεσα στους διάφορους διάβλους που υπάρχουν ε, σε επίπεδο δημοσιονομικό μεταξύ των διαδοτικών ταμείων και των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων παραγωγής χάρη. Και για το ερώτημα τώρα του κυρίου Φερνάντες. Η δική μας εμπειρία είναι ότι τα εργαλεία αυτά τα οποία διαδέχονται τα προηγούμενα εργαλεία έχουν ξεκινήσει με ταχύ ρυθμό, χωρίς καθυστερήσεις, και αυτό αφορά κυρίως το κόσμο και το ορίζον 2020. Τα νέα εργαλεία, τα τελείως νέα, χρειάστηκαν ένα μεγαλύτερο διάστημα προετοιμασίας. Αυτό είναι μια, ένα δίδαγμα το οποίο μπορέσαμε να αντλήσουμε. Αυτό όμως δεν είναι θέμα κανόνων, είναι θέμα τεχνικών συνδικών για να δημιουργήσετε ένα νέο εργαλείο. Πρέπει να προβείτε σε μια ανάλυση της αγοράς εκ των προτέρων, κατά πόσο τα χρηματοπιστωτικά ε, ιδρύματα ενδιαφέρονται για ένα τέτοιο εργαλείο, θέλετε να δημιουργήσετε μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση γύρω από αυτό το εργαλείο και να δημιουργήσετε ζήτηση. Βλέπουμε ότι σε συνολικό επίπεδο, ότι για τα διορθωτικά ταμεία υπολοιπόμαστε αυτού που θα θέλαμε να έχουμε πετύχει σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα. Αυτό είναι μια γενική όμως παρατήρηση, δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών Θεμάτων, DG Radio να διπλασιαστεί η χρήση αυτών των εργαλείων και βάσει των λειτουργικών μας προγραμμάτων στα χαρτιά μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος αλλά σε επίπεδο εφαρμογής Πρέπει να δούμε τι γίνεται, γιατί πολλές φορές είναι μόνο στο τέλος μιας περίοδου προϋπολογισμού που ξεκινούν αυτά τα εργαλεία, οπότε ακόμα βρισκόμαστε στη φάση διαχείρισης των προηγουμένων και τελειώνουν τα προηγούμενα προτού ξεκινήσουν τα επόμενα. Για τη μόχλευση, όπως ε, ρωτήσατε επίσης, αυτό το οποίο βλέπουμε μέχρι στιγμής και θα το δείτε τον Ιούνιο στην έκθεσή μας για την εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων το 2015 τα χρηματοδοτικά εργαλεία προσπαθούν να στοχεύσουν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο μόχλευσης. Καμιά φορά και επέκεινα αυτού του επίπεδου μόχλευσης. Για την προσβασιμότητα στις πληροφορίες, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και πάλι πρέπει να κάνουμε διακρίση δύο επίπεδων. Για τις διαχειριστικές αρχές, είναι φανερό ότι υπάρχει ακόμα ανάγκη τεχνικής αρρωγής που χρειάζονται για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι κανόνες στο τρέχον διάστημα δημοσιονομικών προοπτικών έχουν απλοποιηθεί σε σχέση με, το προηγούμενο, με την προηγούμενη 7 ετία. Η δυσκολία τώρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να ψάξουν κατευθείαν αρρωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουν να ενισχύσουν το μετοχικό κεφάλαιο, τότε μπορούν να πάνε σε ένα, ε, σε ένα ταμείο επενδύσεων, σε ένα ταμείο ε, επενδύσεων με ανάληψη κινδύνου και δεν χρειάζεται να ξέρουν αν αυτό το ταμείο έχει μια υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, αυτό δεν τους μοιάζει. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι Μπορούμε εμεί να υποστηρίξουμε αυτά τα ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Είναι σημαντικό να τα υποστηρίξουμε τα ταμεία αυτά και να έχουν επαρκεί πόρου ώστε να μπορέσουν να δανειοδοτήσουν τι επιχειρήσει αυτέ. Και επίση ή να αυξήσουν το μετοχικό του κεφάλαιο. Και άμα θέλουν ένα δάνειο, τι κάνουν, πηγαίνουν σε μια παραδοσιακή εμπορική τράπεζα. Και εδώ δεν ζητούν άμεσα την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούν κάποιο δάνειο. Και αν υπάρξουν μικρομεσαίε επιχειρήσει οι οποίες έχουν αδυναμίες και εκεί είναι η αστοχία της αγοράς λόγω αυτών των αδυναμιών δεν μπορούν να δανειοδοτηθούν. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει τις τράπεζες να δώσουν αυτή τη δανειοδότηση με την ανάληψη κινδύνου, με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η χρηματοπιστωτική ενδιάμεση, δηλαδή οι τράπεζες <clears throat> έχουν μια πολύ καλή γνώση και συνειδητοποίηση αυτών των δυνατοτήτων. Στι συμφωνίε μα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλου φορεί, εμεί επιμένουμε ιδιαίτερα για το μάρκετινγκ αυτών των εργαλείων και γίνονται συνεχεία εκδηλώσει για να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για την ύπαρξη αυτών των εργαλείων. Αυτό το οποίο είναι για μας πρόκληση είναι να πάμε σε κράτη-μέλη που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Αυτό είναι μια συνολική πρόκληση, δεν είναι θέμα κανόνων γιατί φυσικά οι κανόνε πρέπει να ισχύουν για όλου πρέπει να έχουμε ισότητα ανταγωνισμού, αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να επιτύχουμε την σωστή στόχευση σε κάθε επίπεδο για τη χρήση των εργαλείων αυτών. Υπάρχουν λοιπόν πολλά που μπορούμε να κάνουμε ακόμα σε επίπεδο εφαρμογής και από τις διαχειριστικές αρχές, ώστε να ξεπεράσουμε τα 4-5 κράτη-μέλη που ήδη έχουν όριμο χρηματοπιστωτικό τομέα και ξέρουν να χρησιμοποιούν τα χρηματοπιστωτικά οικονομικά εργαλεία. Κύριε Γουαρδιά Σαβάλ, επίση αναφερθήκατε στο τι προσπαθούμε να κάνουμε για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Θα υπάρξει σύντομα μια πρόταση από την Κομισιόν και θα κάνουμε μια συνδιάσκεψη και για το θέμα αυτό για να τα παρουσιάσουμε. Για τα χρηματοδοτικά εργαλεία κυρίως στοχεύουμε σε μια μεγαλύτερη απλοποίηση σε ό,τι αφορά τα, τις υποχρεώσεις παροχής αναφορών. Έχουμε την υποχρέωση, έχουν υποχρέωση οι επιχειρήσεις να κρατάνε τα αρχεία τους για 7 χρόνια. Η πρακτική της αγοράς είναι μόνο 5 χρόνια. Αν υπάρξει εκεί μια ευθυγράμμιση, αυτό θα κάνει πιο ελκυστικά τα χρηματοδοτικά μας εργαλεία και για τα εργαλεία τα οποία έχουν καθυστερήσει ή έχουν προπορία σε σχέση με το χρονοδιάγραμμά του και εδώ θα κάνουμε κάποιε προτάσει. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι τόσο αλλαγέ στου κανόνε. Αν χρειάζεται θα το κάνουμε. <clears throat> θα κάνουμε κάποιε αλλαγέ, κάποιε προσαρμογέ στα βασικά κείμενα. Αυτό που θέλουμε να εξετάσουμε περισσότερο σε βάθο είναι το εξή. Αν θέλουμε μια διαχειριστική αρχή να χρησιμοποιήσει του κανόνε αυτού για να συμπληρώσει τη χρηματοδότηση ενό εργαλείου, αυτό θεωρητικά είναι δυνατό γιατί είναι κάτι που έχουμε προβλέψει στην ε, ε, βασική πράξη για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά όλα αυτά ακόμα είναι ε, ακόμα λιγάκι ασαφή. Πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η γεφύρωση στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ, λέω Αυτά ήταν λοιπόν οι αρχικές παρατηρήσεις από τον κύριο Μισό σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο. Τώρα έχουμε σε δύο φάσεις την ε, ε ακροάση. Καταρχήν αυτά τα στοιχεία τα οποία τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι αντικείμενο επιμερισμένου ελέγχου και διαχείρισης και αυτών των εργαλείων που βρίσκονται υπό κεντρική διαχείριση. Το πρώτο κομμάτι για την επιμερισμένη διαχείριση ανοίγει με δύο παρεμβάσεις που θα έχει ο καθένας 15 λεπτά στην διάθεσή τους και δίνω το λόγο στην κυρία Πατρίσια Βολίνσκα Κέιβιτς. συγγνώμη εάν δολοφονώ το όνομά σας, είναι υπεύθυνη για την ε, μονάδα της, ε, των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Μπεζεκά, που είναι η Τράπεζα Ανάπτυξης της Πολωνίας. Έχετε το λόγο, κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνουμε σήμερα για τα χρηματοδοτικά μέσα και θα ήθελα καταρχήν να σας πω ποιοι είμαστε, ποια είναι η BGK. Είναι η Εθνική λοιπόν Τράπεζα Προώθησης της Πολωνίας, η οποία ιδρύθηκε το 1924. Ανήκει 100% στο κράτος. Και ε, την χάνει υπό την ε, ε, εποπτεία της Εθνικής Αρχής ε, ε, Εποπτείας των Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων. Βρισκόμαστε στη φάση εφαρμογής μιας σειράς από χρηματοοικονομικά μέσα στην, ε, στο πλαίσιο ε, της ε, ε, περίοδο 2007 έως 2013 και να σας δείξω εδώ ποιο ήταν το σύστημα εδώ που ακολουθήσαμε σε ό,τι αφορά ε, την ε, πρόθεση της ε, κοινωνικής πολιτικής. Να σας πούμε καταρχήν εδώ ότι το σύστημα διαχείρισης στη χώρα μας προβαίνει σε μια διάκριση ανάμεσα στις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και τις αρχές περιφερειακής αυτοδιοίκησης που αναλαμβάνουν δηλαδή τους εκάστοτε ρόλους των αρχών διαχείρισης των λογοταμείων. Στο προηγούμενο λοιπόν ε, πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο που σας ανέφερα στο 2007-2013 είχαμε ένα ε, μεγάλο κομμάτι το οποίο αφορούσε την πολιτική συνοχή, αλλά μόνο το 1% αυτού του συνόλου των κονδυλίων κατευθύνθηκε προς τα χρηματοδοτικά μέσα. Ε, και αυτό το 1% αφορούσε ειδικότερα την υποστήριξη απέναντι στι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την αναζωογόνηση των ε, πόλεων, των αστικών περιοχών, το περιβάλλον και την κοινωνική οικονομία. Ε, η BJK συμμετείχε σε πολλά από αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα ως αρχή διαχείρισης, αλλά να πούμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των κονδυλίων που δεσμεύτηκαν για τα χρηματοδοτικά μέσα εντάχθηκαν στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Είχαμε λοιπόν 16 αρχές περιφερειακής αυτοδιοίκησης στις 16 ε, αντίστοιχες περιοχές της χώρας μας, στα διαμέρισματα η BJK τώρα έπαιξε διαφορετικούς ρόλους στο πλαίσιο της ε, εφαρμογής ε, αυτών των ε, προγραμμάτων. Ήταν για παράδειγμα η αρμόδια αρχή για την καταβολή των πληρωμών σε σχέση με όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία εκτός των αγροτικών ταμείων. Επίσης έπαιξε το ρόλο του χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Τζέσικα σε τρεις διαφορετικές περιοχές και εξακολουθεί να είναι μέχρι και σήμερα ε, η διαχειριστική αρχή για το holding fund, δηλαδή την, ε, το Αμείο Χαρτοφυλακίου, ε, για, συγκεκριμένες, για έξι περιοχές. Επίσης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης της Ανατολικής Πολωνίας και το πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης. Επίσης έχουμε χρηματοδοτήσει ένα ε, πιλωτικό ε, πρόγραμμα χρηματοδότησης με ε, κονδύλια από το ESF και αποτέλεσε ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα γιατί πρόκειται βέβαια για έναν δύσκολο αρκετά τομέα. Και την τελευταία περίοδο η BJK ανέλαβε τα καθήκοντα ε, διαχειριστικής ε, αρχής ε, και πάλι του των κονδυλίων για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το σχετικό Ταμείο Εγγυήσεων της Καινοτόμας Οικονομίας. Επίσης έπαιξε και το ρόλο εφαρμοστικής αρχής σε ό,τι αφορά την υποστήριξη για την αποπληρωμή κονδυλίων τα οποία λήφθηκαν από το ε, ταμείο ε, Τεχνολογικών Επιστώσεων. Τι μάθαμε λοιπόν από αυτή την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ποια ήταν τα διδάγματα που αντλήσαμε. Ε, καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι φτάσαμε σε μια κοινή συμφωνία ότι τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν πραγματικά να εξασφαλίσουν μεγάλα ωφέλη. Γιατί αυτό δεν ήταν προφανές κατά την έναρξη της εφαρμογής ε, ε, της προγραμματικής περίοδου και των χρηματοδοτικών μέσων. Ωστόσο, ε, διαπιστώσαμε ότι με τη χρήση των χρηματοδοτικών ε, μέσων οδηγούμαστε σε καλύτερη ποιότητα των ε, προγραμμάτων και προφανώς μπορούμε ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε και πολύ μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων. Και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο έχουμε περισσότερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και έτσι δίνουμε περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης από την πλευρά της ίδιας της αγοράς. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ανταποκρινόμαστε στις ανεπάρκειες της αγοράς. Καλύπτουμε το χρηματοδοτικό που, κενό που υπάρχει εκεί. Επίσης, ως διαχειριστική αρχή των ε, ταμείων χαρτοφυλακίου σε έξι ε, περιοχές για την πρωτοβουλία Τζέρεμι, είδαμε ότι υπήρξε, ένα πάρα, υπήρχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί ήμασταν ακριβώς ευέλικτοι απέναντι στην κάλυψη των αναγκών για, την, ε, για το χρηματοδοτικό κενό. Και τώρα, το έχουμε ήδη ξεκινήσει με την ε, εφαρμογή του τρίτου ανανόμενου προγράμματος ε, ε, μια συγκεκριμένη περιφέρεια που έχει ξεκινήσει από το 2014. Επίσης να πούμε ότι το νομικό πλαίσιο για τις Δημοσιονομικέ ε, προοπτικέ ήταν αρκετά γενικό, αλλά περιείχε και μια σειρά από οδηγίε, από κατευθυντήρε γραμμέ. Και θα τις αναφέρω συγκεκριμένα αυτές τις ε, οδηγίες που περιλάμβανε, αλλά Ε, βρισκόμαστε ακόμα σε φάση όπου προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα. Και, δηλαδή, το κάναμε και στο παρελθόν και συνεχίζουμε να το κάνουμε γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Εκείνο δηλαδή που είναι σημαντικό είναι να μην αλλάξουμε τα πράγματα, να μην αλλάξουμε το πλαίσιο με τρόπο που να μην δημιουργήσει κινδύνους. Δηλαδή έχουμε δημιουργήσει ένα σταθερό σύστημα, το οποίο τώρα είναι ένα βασικό σύστημα, το, στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε και χωρίς να χρειαστεί να πρέπει να θέσουμε εξ αρχής όλους τους κανόνες. Τώρα να σας αναφέρω ποια ήταν, ε, ποιες ήταν οι θετικές επιτυχές, αν θέλετε της εφαρμογής ε, αυτής της προγραμματικής περίοδου. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες, ε, υπάρχουν κάποιες σαφείς κανονισμοί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνουν τη διακριτική ευκαιρία στα κράτη-μέλη να σχεδιάσουν με τρόπο τέτοιο τα χρηματοδοτικά μέσα τους ώστε να ανταποκρίνονται στις εθνικές ιδιαιτερότητες και να ανταποκρίνονται και στις δυνατότητες χρηματοδότησης γιατί τα ταμεία συνοχής για τα αναπτυξιακά ταμεία ακριβώς δίνουν έμφαση στην περιφερειακή και τοπική διάσταση. Οπότε το σύστημα το ίδιο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις, ε, στα υφιστάμενα ε, κενά ε, της αγοράς, χρηματοδοτικά κενά, τα οποία αφορούν ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και αυτό ειδικότερα όταν αναφερόμαστε στο ζήτημα της ε, ευελιξίας. Δηλαδή διαπιστώσαμε ότι τα όσα μάθαμε στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας δεν χάθηκαν, εφαρμόστηκαν. Και το επίσης θετικό, ένα ακόμα θετικό ε, στοιχείο ήταν ότι η καθοδήγηση, το guidance είχε δημοσιευθεί πριν από την έναρξη της εφαρμογής. Όχι πάντοτε, αλλά συνέβη, έγινε ε, κάποιες φορές. Κάτι ακόμα θετικό ήταν ότι όταν υπήρχαν οδηγίες, προσπαθούσαν απλώς να ερμηνεύσουν, να αποσαφηνίσουν τους υφιστάμενους κανονισμούς. Δεν προσπαθούσαν δηλαδή να τους καταστήσουν πιο αυστηρούς. Επίσης, να πω ότι έχουμε, είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία ε, μεταξύ των ε, χρηματοδοτικών διαμεσολαβητών και ε, τις, ε, τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως βέβαια και, των, ε, και μεταξύ μόν και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο ακριβώς της εκταμίευσης των κονδυλίων. Όμως να σας πω τώρα τι δεν λειτουργήσε τόσο καλά. Καταρχήν είχαμε υπερβολικά περιοριστικούς και περίπλοκους κανόνες για την εφαρμογή Επίσης, οι οδηγίες που δημοσιεύονταν για τα εν λόγω project είτε δημοσιεύονταν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, δηλαδή καστερημένα, ή ακόμα χειρότερα κατά την ε, εφαρμογή ε, των εν project. Ε, είδαμε ότι συχνά εστιαζόταν σε πολύ τεχνικές λεπτομέρειες. Ε, αλλά δεν είναι δυνατόν να αλλάζει κανείς του κανόνες του παιχνιδιού όταν ήδη έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Οπότε θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό εδώ. Γιατί σε αυτή την περίπτωση κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τελικά ε, τι να περιμένει κατά την έναρξη του προγράμματος και έτσι το αποτέλεσμα βέβαια δεν είναι τόσο ε, πρόσδεκτο. Κάτι ακόμα τώρα που δεν ήταν ε, πολύ θετικό ήταν ε, το γεγονός ότι το σύστημα σχεδιάστηκε με μια ε, δομή, αν θέλετε, από τα πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή από το κεντρικό, αν θέλετε, επίπεδο προς το κατώτερο. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα θετικό για τους δικαιούχους. Από εκεί και μετά ποιε είναι οι προκλήσεις. Να πούμε ότι ένας σοφός άνθρωπος ε, είπε κάποτε ότι η ε, τελειότητα δεν επιτυχάνεται όταν δεν υπάρχει πλέον ε, κάτι να προσθέσουμε στο, στο αποτέλεσμα, αλλά επιτυχάνεται όταν δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μπορούμε να αφαιρέσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε λοιπόν, να σας πω τι μπορούμε να έχουμε ε, την πρόκληση για την τρέχουσα τώρα ε, προγραμματική περίοδο. Υπάρχουν κάποιες, κάποια βεβαιότητα καταρχήν σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο, ειδικότερα και, το, και, τα, και τις διατάξεις και του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, του CPR. Ε, και αναρωτιόμαστε κατά πόσο με βάση όλες αυτές τις διατάξεις τελικά απομένει κάποια ευελιξία την οποία να παρέχει το σύστημα. Και νομίζω πως αυτό θα αποτελέσει και αντικείμενο των συζητήσεων μας και σήμερα και στο μέλλον. Μετά, δημόσιες συμβάσεις και οι κανόνες που διαπούν τις δημόσιες συμβάσεις. Για παράδειγμα, η διαδικασία επιλογής των, εφαρμοστικών, των φορέων εφαρμογής ο, ο τρόπος που έχει σχεδιαστεί δεν εξυπηρετεί τον στόχο, δηλαδή να έχουμε μια ευέλικτη διαδικασία η οποία θα προσαρμόζεται στις ανάγκες αγοράς και του συστήματος. Επίσης, είδαμε ότι έχουμε πάρα πολύ σύγχρονους ε, περιορισμένους ε, ε, κανόνες στο πλαίσιο της, του κανονισμού και λίγες οδηγίες, οδηγίες περαιτέρω, περιορισμένη δηλαδή καθοδήγηση. Ε, αλλά τώρα που ξεκινούμε την προγραμματική περίοδο, την νέα προγραμματική περίοδο, ήδη έχουν αυξηθεί σε 11 ο αριθμός των οδηγιών που έχουμε λάβει. Και επίσης ε, ε, εκείνο που είναι θετικό είναι ότι λάβαμε το πράσινο φως για να δημιουργήσουμε ε, τις δικές μας οδηγίες οι οποίες θα προσανατολίζονται στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι κανόνες που ίσχυαν μέχρι τώρα δεν εμ, το σύστημα, το ευέλικτο σύστημα που έχουμε δημιουργήσει τώρα και θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να καταστρέψουμε τα όσα έχουμε μάθει μέχρι τώρα, να τα αγνοήσουμε. Άρα λοιπόν αποτελεί ιδιαίτερα μεγάλη πρόκληση η ευελιξία. Μπορούμε όμως να την επιτύχουμε, ναι, με κανόνες εφαρμογής, αλλά ε, με κανόνες οι οποίοι ταυτόχρονα θα λαμβάνουν υπόψη την ευελιξία η οποία χρειάζεται ε, για την ε, αγορά. και θα επιτρέπουν μια δημιουργική προσέγγιση και από τους ε, ε, εταίρους χρηματοδοτικούς διαμεσολαβητές. Ειδικότερα δε εάν θέλουμε να ανοίξουμε ακριβώς τους διάβλους, δηλαδή να έχουμε περισσότερους συμμετέχοντες ως χρηματοδότες. Τώρα, στο επίπεδο της ε, πολιτικής συνοχής για την, προγραμματική, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο έχουμε προβλέψει γύρω στα 4 ε, δις ευρώ για την εξάντια ανάλυση, δηλαδή ένα τετραπλάσιο ε, ποσό σε σύγκριση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Ε, θέλουμε λοιπόν να είμαστε παρόντες και να δημιουργήσουμε ή ε, να έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα προσαρμοσμένο ε, σύστημα σε διάφορες ε, περιοχές, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Τι θέλουμε να επιτύχουμε με όλα αυτά. Δεν θέλουμε να έχουμε πάρα πολύ λεπτομερείς οδηγίες. Για παράδειγμα, το ζήτημα του accountability, της ευθύνης και της διαφάνειας είναι ζητήματα τα οποία μπορούμε να τα διασφαλίσουμε χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως αυτοί ίσχυαν ε, για τις ε, ενισχύσει. Δηλαδή να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τις ενισχύσει, ε, που ίσχυαν για τις ενισχύσεις να ισχύουν και για τα χρηματοδοτικά μέσα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που μας δείχνει ότι εκείνο ε, που δημιουργήθηκε στην αγορά κατά τα τελευταία 15 χρόνια δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα, για παράδειγμα, δίνοντας εγγυήσει στους ε, ε, δικαιούχους από, τον, από την αγορά. Κάτι, ένα τέτοιο ρόλο δεν χρειάζεται να το παίξουμε, οπότε γιατί να εφαρμόσουμε αυτούς τους παλαιότερους κανόνες για ε, τα μία τώρα σε αυτή την περίοδο και από εκεί και μετά εκείνο που είναι σημαντικό είναι να μειώσουμε το διοικητικό άχθος, δηλαδή να μην, ε, έχουμε, να μην χρειάζεται να εφαρμόζουμε μία σειρά από πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την εξάντια αξιολόγηση, όταν οι διαχειριστικές αρχές καλούνται να ε, προβαίνουν σε εξάντια ανάλυση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Για παράδειγμα, όταν προβλέπονται τρει ε, τέτοιου είδου εξάντε αναλύσει, για παράδειγμα για τι εγγυήσει, για τα δάνεια και ούτω καθεξή, ε, δεν νομίζουμε πω κάτι τέτοιο έχει χρησιμότητα. Είναι υπερβολικό. Οπότε θα πρέπει λίγο να εξετάσουμε πώ μπορούμε να πλουστεύσουμε τη διαδικασία και να αποφύγουμε τη δημιουργία περισσότερου διοικητικού φόρτου εργασία. Γιατί σήμερα ήδη υπάρχει τέτοιο φόρτο. Σα ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα γιατί τα συμπεράσματα που θα βγουν από αυτήν την ε, συζήτηση και εκθέσεις που θα ακολουθήσουν θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και στο πλαίσιο της ε, επόμενης ε, προγραμματικής περίοδου. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου και χαιρόμαστε για αυτά που είπατε. Τονίσατε την ανάγκη της απλοποίησης και την άρση του άχθους που προέρχεται από τις υπερβολικές αξιολογήσεις κτλ. Ο κύριος τώρα Αλεξάντερ Μπάρτελ, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομίας και Ενέργειας Ζεδεάς και επικεφαλής της ομάδος ε, δράσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην οργάνωση των Ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Έχετε το λόγο κύριε Μπάρτελ. Oh, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω εδώ στις Βρυξέλλες και να συζητήσω μαζί σας για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από τη δική μας ε, οπτική γωνία και ιδίως τη γερμανική οπτική γωνία μπορώ να σας δώσω ορισμένα στοιχεία. Εμείς είμαστε ε, μια ένωση περίπου ενός εκατομμυρίων επιχειρήσεων με πέντε ε, εκατομμύρια εργαζόμενους, άρα περίπου 5 άτομα κατά επιχείρηση. 80% των επιχειρήσεων της Γερμανίας έχουν ε, μικρότερο τσίρο από ένα εκατομμύριο και λιγότερους από, από 40 εργαζόμενους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η χρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων και εμείς είμαστε πάντα ε, υπέρ του να υπάρξει μια διεύρυνση της δυνατότητας των χρηματοδοτήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι μόνο από τις κλασικές ε, μορφές διαμεσολόβησης. Ευτυχώς η Γερμανία έχει ένα οργανωμένο σύστημα τοπικών ε, φορέων όπως είναι τα ταμιευτήρια σε τοπικό επίπεδο που καλύπτουν πάνω από 84% των συνολικών αναγκών των επιχειρήσεων. Και επίσης έχουμε και τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία κατευθύνονται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως για να μπορέσουν όλα αυτά τα ιδρύματα να φέρουν σε πέρα στο έργο τους όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να επιτύχουν το στόχο τους, τότε δημιουργείται πολλές φορές και ένα χάσμα. Και δημιουργούνται και κίνδυνοι που θέτουν ένα αμφιβόλο την ε, λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών και την δυνατότητα να μπορούν να προχωρήσουν τη δραστηριότητά τους γιατί μόνο εν μέρη μπορεί να εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους. <clears throat> Ένας από τους ε, βασικούς λόγους για τους οποίους θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι έχουν αγωνιστεί στο να υπάρχει ένας ε, συντελεστής διόρθωσης στην ομάδα 1 αυτό είναι και ένας ε, βασικός παράγων ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την διαθεσιμότητα των κονδυλίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και έχουμε διαπιστώσει ενδιαμέσως ότι ο παράγων αυτός διόρθωσης μπορεί να λειτουργήσει και φυσικά υπόκειται πάντα σε μια διαδικασία ελέγχου σε δύο επίπεδα. Πιστεύουμε ότι είναι φυσικά απαραίτητο να συνεχίσει και στο μέλλον μια συνεχής αξιολόγηση του παράγοντος του συντελεστή αυτού <clears throat> διόρθωσης. Κάθε δύο χρόνια θα πρέπει να έρχεται και πάλι σε εξέταση αυτός ο παράγον για τις πιο μακροχρόνιες πιστώσεις οι οποίες δίνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τι ακόμα χρειαζόμαστε, ή για ποιο λόγο και τι δεν χρειαζόμαστε από τις ε, χρηματοδοτήσεις αυτές είναι κυρίως οι υπερβολικές στατιστικές απαιτήσει που ζητούνται σε μας από τις ε, αρχές και την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και εδώ πάλι θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι με τις ακροάσεις αυτές έχουμε την δυνατότητα να εκφράσουμε την απόψή μας και να διορθωθούν ορισμένες ελλείψεις που υπάρχουν και που υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις για ένα κονδύλιο 20-25 ευρώ πολλές φορές να δώσουν ένα όριμαγδό πληροφοριών που δεν ε, έχουν καμία αξία για, τις, ε, τα πιστοτικά μας ιδρύματα και που φυσικά οδηγούν και σε περαιτέρω επιβάρυνση για τα ταμιευτήρια και τα πιστοτικά ιδρύματά μας. Και κάτι άλλο που χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο στην Ευρώπη. Μπορώ να επιθυμήσω αυτό που είχε πει ο κύριος Καράς στην ε, παρουσίαση της έκθεσης πρωτοβουλίας τους. Χρειάζεται να υπάρξει μια διαφοροποίηση του τομέα χρηματοδότησης και φυσικά να μην υπάρχει μονάχα η ανάγκη πρόσβασης σε τραπεζικά κονδύλια, να υπάρχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής για τις επιχειρήσεις, κάτι το οποίο να έρχεται σε καλύτερη προσαρμογή με τις ε, επιχειρήσεις μας που δεν είναι πάντα οι περισσότερες επιχειρήσεις, βιοτεχνικές επιχειρήσεις δεν είναι στα ίδια επίπεδα με τις μεγάλες επιχειρήσεις που χρειάζονται κεφάλαια. Έχουμε εδώ τις ε, τράπεζες οι οποίες ε, πολλές φορές μπορούν να παράσχουν προγράμματα αναπτυξιακού χαρακτήρα. Αλλά αυτά τα προγράμματα δεν πρέπει να έχουν μεταξύ τους ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Παραδείγματο χάρη έχουμε το πρόγραμμα, το σχέδιο ΕΦΣΥ και έχουν δοθεί δάνεια στην ε, στις κάτω χώρες δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Γιατί όμως και στην περίπτωση της ε, Γερμανίας, όπου δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Δεν πρόκειται για χώρες οι οποίες χωρίζονται από τις Άλπεις, αλλά απλώς από ένα ποταμό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πιο συνολική μορφή συντονισμού που να υπερβαίνει τα εθνικά ε, όρια σε σχέση με το πώς τα ευρωπαϊκά όργανα και τα χρηματοπιστωτικά όργανα δίνουν βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ. Merci, monsieur, pour... Σας ευχαριστώ πολύ για την άποψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό το οποίο χρειάζονται οι επιχειρήσεις αυτές για την αναπτυξή τους δεν είναι τόσο τα εργαλεία όσο οι πιστώσεις. και ή δυνατόν να μην είναι τόσο σφιχτός ο κορσές στον οποίο τις υποχρεώνουν και όχι μια πολυπληθώρα στατιστικών στοιχείων που θα πρέπει να αναφέρουν. Έρχομαι τώρα στις δύο υπεύθυνες ακρόασεις. Έχετε να θέσετε κάποια ερωτήματα, κυρία ε, Ριάντα, κυρία Γουάρδια Σαβάλ, κυρία Σαρβαμά. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Σαρβαμά ένα ερώτημα και εν μέρη σχόλιο. Για την κυρία Βόνης Καμπαρκέβιτς. Εκεί που λέγατε για τα συμπεράσματα του περιοδου 2007-2013, εκεί δεν κατάλαβα τι γινόταν. Μήπως μπορείτε να διευκρινίσετε ή κάπως να επικρατείτε. γιατί και τα δυτικά και τα αρνητικά εδώ είναι σχεδόν ταυτόσιμα. Δηλαδή το ένα απέδωσε και το ίδιο πράγμα δεν απέδωσε, που δεν σας πρόσεξε αρκετά. Θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα, οπότε χρειάζονται και συγκεκριμένα παραδείγματα από συγκεκριμένα προγράμματα, έργα και να δούμε ε, τι, τι γίνεται και να δούμε αν υπάρχει αντίφαση. Και τώρα, κάποια άλλη ερώτηση, κάποιο που δεν είναι ειδικό. Εάν κατάλαβα καλά, όπω είπε και ο πρόεδρο. απλούστευση των κανόνων. Συμφωνώ πάνω σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι είπατε δεν σας πάρα πολύ αυτή η αντιμετώπιση εξάντε εγώ όμως νομίζω ότι η τάση είναι όλο ένα και πιο ε, σημαντική μια τέτοια αντιμετώπιση και όχι το αντίθετο. εντάξει, υπάρχει διαφορά σε κάποιε πολιτικέ ομάδε, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα προ εκείνη την κατεύθυνση πάνε. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζει κανεί εκ των προτέρων ε, πού θα διαθέσει τα χρήματα των προλογουμένων και αν θα αποδώσουν. Οπότε και εδώ θα πρέπει να ε, ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα για να έχουμε απλούστευση και αποτελεσματικότητα. Merci, Monsieur Olbricht. Κύριος Olbricht. I think in the, in the framework of our debate on MFF revision, για την προσπάθεια διόρεσες του πλούς πλαισίου. Είναι σημαντικό να λάβει υπόψη και αυτά που λέμε τώρα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. σε είναι και τον Σαρβαμά. Προκεί κάτι που δεν πάει καλά. Βρισκόμαστε στη μέση της ζωής του πολιτού πλαισίου. Μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα. Να αλλάξουμε τις καθεντήριες για το επόμενο πολιτές πλαίσιο μετά το 2020. Να αλλάξουμε τώρα, ας πούμε, τις έντες γραμμές, αλλά αν υπερβολικά πολλές. και αν η εκ των προτέρων που είναι κάτι το σωστό υπάρχει. Αλλά από ό,τι κατάλαβα. Έχουμε τώρα πολλαπλασιαζόμενες τέτοιες ε, ε, τέτοια αντιμετώπιση. Επομένως, θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση. Αλλά θα πρέπει με το 2020 να το κάνουμε αυτό ή να το αλλάξουμε εδώ και τώρα. Ο κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ πολύ. If I could ask a question. Στο συγγνώμη μπορώ να θέσω ένα ερώτημα. Ποιος μικρόφωνο, Πρόεδρος. I'm sorry. Not now, not now. Oui, vous aurez la parole tout à l'heure, mais je venais de donner la parole à M. Rubig. Θα σα δώσω το λόγο αμέσως, αλλά προηγουμένω τον κύριο Ρίμπιχ. Κύριε Ρίμπιχ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στον κανονισμό 651 του 2014, όπου αναφέρονται τα χρηματοδοτικά μέσα και ε, στην, ε, στην περίπτωση όπου ενδέχεται να μην υπάρχουν τα ε, απαραίτητα κονδύλια, για παράδειγμα επειδή οι επενδύσεις ε, έχουν απορροφηθεί ε, σε συγκεκριμένα άλλα ε, project, οπότε εκείνο που τελικά ο στόχος είναι θέλουμε να βελτιώσουμε την χρηματοοικονομική κατάσταση. Οπότε, εάν κάποιες επιχειρήσεις αντιμετωπίσουν προβλήματα, σήμερα τουλάχιστον δεν έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση, Ακριβώ επειδή δεν προβλέπεται αυτό ο μηχανισμό πλέον. Οπότε, στο πλαίσιο των τοποποιήσεων προβλέπεται να κάνετε, πιστεύετε ότι ε, θα μπορέσει να ληφθεί και αυτό υπόψη. Γιατί προφανώ, προφανώς η ρευστότητα των επιχειρήσεων είναι ένας πολύ σημαντικό παράγοντας και δεν καλύπτεται επαρκώς και αναφέρεται επανειλημμένα και το ε, κεφάλαιο κινδύνου του Risk Capital από την Επιτροπή και πράγματι θα πρέπει να το υποστηρίξουμε ούτως ώστε να έχουμε περισσότερες επενδύσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε καινοτομίε. Χωρίς να το κάνουμε αυτό δεν θα επιτύχουμε τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οπότε θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο σαφείς ως προς το στο τι θέλουμε να επιτύχουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριος Μάη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω ε, ένα σύντομο ερώτημα στον άνθρωπο που με μίλησε πρώτος. Νομίζω πως αυτό το ζήτημα αφορά ε, όλες, ε, όλα τα κράτη-μέλη, αλλά ειδικότερα και την Ιρλανδία. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά ε, θα υπάρξει ε, μια συνεργασία μεταξύ της, ε, του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Ταμείου, Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και της αρμόδιας τράπεζας προώθησης της Ιρλανδίας. Μόνο με αυτό το μοντέλο θα λειτουργήσει η διάθεση αυτών των μέσων. Άλλα ερωτήματα δεν βλέπω να υπάρχουν. Και εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Μήπως το να επιζητούμε να θέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει καλύπτει 28 κράτη-μέλη στην υπηρεσία των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι η πεμπτουσία του αποκεντρωμένου τοπικού οικονομικού ιστού. Μήπως στην περίπτωση αυτή θα πρέπει αυτή η χρηματοδότηση που αυτή τη στιγμή γίνεται από πιστοτικά ιδρύματα να βελτιωθεί. Πώς μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα αυτά φτάνουν κατευθείαν στις επιχειρήσεις. Εγώ δεν ξέρω να υπάρχουν επιχειρήσεις μικρομεσαίες που να είναι βιώσιμες και οι οποίες να μην βρουν χρηματοδότηση. Πολλές φορές οι δυσκολίες βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ότι τα κατημέρια δεν έχουν κάνει ακόμα τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να εξασφαλίσουν την δυνατότητα βιωσιμότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ο φόβος μου λοιπόν είναι ότι όταν ξεκινούμε μια επιχείρηση από το ευρωπαϊκό επίπεδο θα συνοδεύεται πάντα με μια πολυπληθώρα κανονισμών, νομικών βάσεων, εξετάσεων εκ των προτέρων. Θέλουμε κίνδυνο ή δεν θέλουμε κίνδυνο. Όλα αυτά δεν είναι εύκολο να τα ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη για να προχωρήσουμε και να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Θέλετε να απαντήσετε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου στα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν η κυρία ε, πρώτα. Συμπαθάτε μου η διαφορά μεταξύ του προηγουμένου και του τώρα ισχύοντος πολιτικού πλαισίου είναι το εξή ότι πριν δεν είχαμε τόσες διατάξεις στο νομικό πλαίσιο. Οπότε και αναπτύχθηκε αυτό το σύστημα παντού. Ας πούμε στην Πολωνία έχουμε ένα σύστημα διαφοροποιημένο πολλαπλά επί τη βάση των ε, περιφερειακών διοικητικών μονάδων και περιφερειών και οι δικαιούχοι δεν είναι εμπορικές τράπεζες. Οπότε μας δώσουν το πράσινο φως του ώστε να φτιάξουμε αυτό το σύστημα και να υλοποιήσουμε αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Ο στόχος μας ήταν να άρουμε τα κενά της λειτουργίας τη αγοράς. Οπότε, αντίσαμε και πέσει συμπεράσματα. Μάθαμε το μαθήμα μας γιατί είναι σημερινή τωρινή περίοδο. Αλλά ακόμα ε, εξελίσσεται το ισχύον σύστημα και γι' αυτό και έχουμε ε, θεσπίσει και νομοθεσία αλλά και κατευθυντήρες. 11 κατευθυντήρες έχουμε μέχρι τώρα εκδώσει για να καλύψουμε ε, κάποια προβλήματα τεχνικά και λειτουργικά τα οποία πολλές φορές ε, δεν, δεν, δεν συνάδουν, δεν έχουν συνάδει με το σύστημα το οποίο προίσχυε και ισχύει. Και προχωράμε. Κάτι φτιάξαμε καινούργια και γι' αυτό και έχουμε τους ενδιάμεσους. Είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δεν είναι εμπορικές τράπεζες. Είναι κάποια ταμεία για δανεισμό, ε, εγγυητικά, ιδρύματα ε, που κινούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οπότε στην τωρινή σημερινή περίοδο θέλουμε να υπάρχει ένα, ας το πούμε, στάνταρ σύστημα. Και αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Ότι η πολυνομία είναι πρόβλημα για την εφαρμογή ε, και χρησιμοποίηση αυτών των εργαλείων χρηματοδότησης. Α, το ίδιο και στην πολιτική συνοχή, οπότε τα διευθυντικά ταμεία έπρεπε να χρησιμοποιηθούν και να επιστρατευτούν όχι για να διώξουν τον ιδιωτικό τομέα, αλλά ε, για να συνδράμουν τα πιο προβληματικά έργα και προγράμματα. άμα λειτουργούσαν 100% οι ιδιωτικέ προσπάθειε δεν θα χρειαζόντουσαν αυτά τα μέσα. Τώρα όμω χρειάζονται. Και αν το σύστημα αυτό το εξελίξουμε και παραέχουμε πολλές αξιολογήσεις των προτέρων, δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε ε, του στόχου, μας, δηλαδή την λύση των τη αγορά. γιατί είδαμε ότι οι περισσότερε αρχέ. Ε, έχουν συμβληθεί με συμβούλους για να γίνει αυτή η εξάντε ε, αξιολόγηση. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν αυτές οι εξάντε αναλύσεις. Οπότε και οι διοικητικές αρχές θα έπρεπε να προσαρμόσουν τις αναλύσεις τους στις κατευθυντήριες που έχουν εκδοθεί. Ωραία, σωστό αυτό. Αλλά στη συνέχεια ε, διαπιστώθηκε ότι έχει ημερομηνία σε αυτή η τακτική. Δηλαδή τι διαπραγματεύσει του κάθε λειτουργικού προγράμματος, η δε κατάσταση στην αγορά αλλάζει ταχύτητα. Οπότε και αυτό το είδαμε την περίοδο 8, 9, 10, 11 μέχρι και 12. Οπότε είχαμε τα λειτουργικά προγράμματα και είχαμε κάποιους ε, δείκτες από τη στρατηγική της Λισαβόνας. Οπότε και θα έπρεπε να μετέλθουν, να χρησιμοποιήσουν τους αυτούς τους δείκτες και το 2008 είδαμε τα πρώτα αποτέλεσματα της ε, οικονομικής κρίσης και άλλαξε κατά στην αγορά ε, ακριβώς γιατί το σύστημα ήταν ευέλικτο οπότε και εμείς μπορούσαμε να ρίξουμε στην αγορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία ήταν κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των προβλημάτων της αγοράς. Χρειαζόταν το η εξάντια ανάλυση. Αλλά, εάν μηχανισμό θα θεσπιστούν ακόμα περισσότερες αξιολογίες εξάντε, πριν από κάθε φάση, από κάθε βήμα, τότε αυτό θα είναι καλό για τη δουλειά των συμβούλων, αλλά δεν θα είναι σωστό για την πολιτική των ε, χρηματοδοτικών εργαλείων. Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Προσοχή στη χρήση αυτών των αναλύσεων εξάντα. Και ένα από τους λόγους των καθυστερήσεων ε, εφαρμογή στην ε, τωρινή περίοδο είναι η αβεβαιότητα. Γιατί οι διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών προγραμμάτων στην χώρα δεν έχουν ολοκληρώσει την ε, διαδικασία των εξάντε αναλύσεων. Merci, Σας ευχαριστώ πολύ. Από, την, ε, από αυτά που είπατε νομίζω ότι δεν λειτουργεί το σύστημα. Δίνω το λόγο. Στον κύριο Κέρο Μουσό, λέει ο πρόεδρος, αλλά προηγουμένως τον κύριο Μπαρτέλ. Κύριε Μπαρτέλ, έχετε το λόγο. Θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια μετά από τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν. Επειδή δεν μου απευθύνθηκε κάποιο άμεσο ερώτημα, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση απλώς. Στην πράξη, τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να αντισταθμίσουν κάπως τις αστοχίες της αγοράς. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα χρηματοδότησης, δεν πρέπει εμείς φυσικά να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις, ε, αυτά τα, τα εργαλεία για να αντισταθμίσουν μια την οργάνωση αυτή των χρηματαγορών που έχουν σαν στόχο να εξασφαλίσουν και τη σταθερότητα των πιστοτικών αγορών και τα οποία βασίζονται στην, ε, ε, στο αξιόχρεο των επιχειρήσεων. Και σας πενθυμίζω για αυτό το οποίο γίνεται στην ε, Επιτροπή της Βασιλείας για μια νέα διαμόρφωση των κριτηρίων ε, κινδύνου σε ό,τι αφορά χάρη τα, τα κτίρια και άλλα στοιχεία ενεργητικού που έχουν σημασία πολλές φορές για τη χρηματοδότηση μιας επιχείρησης. Και πιστεύω ότι και η συζητήσει στο Κοινοβούλιο για το μέλλον του παράγοντα ε, διόρθωσης θα έχουν μεγάλη σημασία. Alors, avant de και πρώτο περάσω στη δεύτερη φάση, κύριε Κερομισό, εσείς που αναφερθήκατε στο ρυθμιστικό πλαίσιο, μετά από αυτά που ακούσατε από την κυρία Μπάρκεβιτς και από τον κύριο Μπάρτελ, έχετε την εντύπωση ότι τα εργαλεία σας είναι πράγματι λειτουργικά ή όχι και υπάρχει ζήτηση για αυτά τα εργαλεία. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση για αυτά τα εργαλεία στο μέλλον ή όχι. Στο τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ναι, θα ήθελα να πω συντριπτικά ναι. Χάρη και στο σχέδιο Γιούν και το σχέδιο Εύση έχουμε καταφέρει <clears throat> να ανταποκριθούμε στην τεράστια ζήτηση που υπήρξε για ένα από αυτά τα εργαλεία ένα είδος εργαλείου που είναι οι εγγύσει για τα τραπεζικά δάνεια προς τις μικρομεσαίες. Έχουμε πολλά εργαλεία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες στο πρόγραμμα COSME, Horizon 2020 και επίσης και για τις πολιτιστικές επιχειρήσεις. Έχουμε λοιπόν εργαλεία που βοηθούν τις τράπεζες, μας ζητάει η τράπεζα μια υποστήριξη και δημιουργούμε εν μια εγγύηση για ένα χαρτοφυλάκιο δανείων που θα δώσει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Το, το σχέδιο Εύση μας επέτρεψε να ανταποκριθούμε σε αυτή την ε, <clears throat> ζήτηση. Και εδώ δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα γίνουν μεγάλες τροποποιήσεις στην ενδιάμεση αναθεώρηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Αλλά το Εύση μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Τώρα, Φυσικά είναι μια επιτυχία το ότι έχουμε επιτύχει τη ζήτηση αυτή. Το <clears throat> επόμενο πρόβλημα τώρα είναι, ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την προσθετικότητα. Μα αυτό είναι το πραγματικό θέμα, λέει ο κύριος Σάτου, γιατί άμα δώσετε στους τραπεζίτες μία εγγύηση, εγώ στοιχηματίζω ότι θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση για δάνεια. Σημαίνει αυτό ότι υπάρχει μια προσθέμενη αξία ή ότι βολεύει πολλούς αυτή η παροχή εγγύσεων. Τόσο ενιολογικά όσο και σε επίπεδο λογιστικού ελέγχου θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να έχουμε μια σωστή ισορροπία. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει αρκετά καλά γιατί ζητάμε από τις τράπεζες να μας δώσουν αποδεικτικά στοιχεία και εφαρμόζουμε μία σειρά από κανόνες για να είμαστε σχετικά πεπισμένοι ότι τα δάνεια αυτά είναι δάνεια τα οποία δεν θα δίνανε οι τράπεζες χωρίς τις εγγύησεις. Τόσο σε ό,τι αφορά την, τους δικαιούχους και σε ό,τι αφορά και τον όγκο των κονδυλίων. Όπως σας έλεγα όμως στην αρχή δεν υπάρχει κάποια μαθηματική φόρμουλα για τα θέματα αυτά. Αυτά είναι πάντα κάτι το οποίο το κάνουμε, το δοκιμάζουμε και υπάρχει μια συνεχής διόρθωση. Αν θέλετε λοιπόν μπορούμε να κλείσουμε αυτή το, αυτό το πρώτο τμήμα και θα περάσουμε στο θέμα της ε, ε κεντρικής διαχείρισης με πρώτο ε, παρεμβαίνοντα το Κριστιαν Ντουμπαρί, ο οποίος είναι αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις στην BPI Γαλλία. Είναι μια θεατρική εταιρεία η BPI του Ταμείου ε, Υποθηκών και παρα, και Παρακαταθηκών στην Γαλλία και έχει τον λόγο για 15 λεπτά κ. Διμπάρη. so my presentation... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην δική μου ε, παρουσίαση θα σας ε, παρουσιάσω ε, τη δική μας εμπειρία με τα κεντρικά χρηματοδοτικά μέσα. Καταρχήν να σας αναφερθώ εν συντομία στην BPI France. Όπως είπατε είμαστε μια θηγατρική της SDC και ε, του Δημοσίου της ε, Γαλλίας ε, ιδρυθήκαμε το 2013 από την συγχώνευση ήδη υφιστάμενων φορέων. Έχουμε έξι τομείς δραστηριότητας, εγγυήσεις, δάνεια, καινοτομία, τα επωνομαζόμενα funds of funds, οι επενδύσεις μικρών κεφαλαίων και οι επενδύσεις μεγάλων και ε, μεσαίων και μεγαλύτερων ε, κεφαλών και υποστηρίζουμε άμεσα τις επιχειρήσεις είτε μέσω χρηματοδότησης ε, δανείων είτε μέσω συμμετοχικών δανείων equity. Τώρα, η δική μας προσέγγιση είναι business friendly, δηλαδή να είμαστε εύκολα προσβάσιμοι, θετικοί, αισιόδοξοι και προσπαθούμε να βέβαια να αυτές, αυτή η προσέγγιση και αυτή η η νοοτροπία μας αν θέλετε να ευθυγραμμίζεται ταυτόχρονα βέβαια και με τα ε, ευρωπαϊκά ταμεία και νομίζω πως το καταφέρνουμε. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος ε, ως NPB, ως ε, δηλαδή Εθνική Τραπέζα Πρόθεσης, ε, ο, φίλος Νεομινίκ θα προβεί σε μια ευρύτερη παρουσίαση, αν θέλετε, του ρόλου των NPB σε σχέση με τα χρηματοδοτικά μέσα, αλλά επιτρέψτε μου και εμένα πολύ σύντομα να αναφερθώ σε μια ανακοίνωση του 2015 σε σχέση με το ρόλο των εθνικών τραπεζών προώθησης για την ε, πρόθεση της ανάπτυξης στην ε, Ευρώπη όπου τονίστηκε ο ρόλος που μπορούν να παίξουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα ENPPs ε, για την πρόθεση της ανάπτυξης. Η ανακοίνωση εκείνη προέβλεπε μάλιστα έναν, υπεριείχε έναν αρκετά ευρύ διαστατικό ορισμό των NPPs και των αναπτυξιακών προγραμμάτων, επενδυτικών προγραμμάτων και ε, αναφέρθηκε εκεί από την ε, Επιτροπή ε, και η εμπειρογνωμοσύνη που έχουν οι NPBs ακριβώς λόγω της εστίασης στο τοπικό επίπεδο και επίσης αναφέρεται ότι λιένουν, ακριβώς προλιένουν το δρόμο προς μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ NPBs και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ρόλο των NPB σε σχέση με τα χρηματοδοτικά μέσα να σας κάνουμε μια παρουσίαση από τη δική μας ε, ε, οπτική γωνία. Ε, δηλαδή, ποια είναι τα χρηματοδοτικά μέσα σε σύγκριση με τα με τις ενισχύσεις. Καταρχήν δεν έχουν τόσο μεγάλο κίνδυνο του να, υπάρξουν, να υπάρχει κατάχρηση, δηλαδή, δηλαδή να αξιοποιούνται από άτομα τα οποία δεν προβαίνουν στις κατάλληλες επενδύσεις. Επίσης έχουν υψηλότερο αντίκτυπο ε, στην, ε, ε, στην αγορά από ό,τι ενισχύσει γιατί ακριβώς μοχλεύουν ιδιωτικό κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση και επίσης δίνουμε αυτόν τον τρόπο κίνητρο στον δικαιούχο να αξιοποιήσει με τον πιο ορθολογικό τρόπο τα σχετικά κονδύλια και επίσης τα χρήματα τα οποία εξοφλούνται στη συνέχεια μπορούν να επανεπενδυθούν και αυτό δημιουργεί ακριβώς ένα πολλαπλασιαστικό αν θέλετε αποτέλεσμα αυτό το multiplier effect. Όμως ταυτόχρονα οι ενισχύσεις ε, ε, παραμένουν απαραίτητες σε ορισμένους τομείς παρόλα αυτά, παρότι δηλαδή είναι καλύτερα τα χρηματοδοτικά μέσα και αυτό σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς όπου τα χρηματοδοτικά δηλαδή μέσα δεν μπορούν να επιλύσουν όλες τις ανάγκες χρηματοδότησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων, είπαμε ότι ο ρόλος των NPBs είναι πάρα πολύ σημαντικός. Όχι, ε, όχι μόνο ε, ως ο κύριος δικαιούχος αυτών των ε, εργαλείων, χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η αρχή η οποία μπορεί να συνενώσει, αν θέλετε, να συντονίσει τις διάφορες αρχές του, ώστε να μπορέσει να προσελκύσει και ε, το, τα ιδιωτικά κονδύλια, τα ιδιωτικά κεφάλαια αυτή, ε, εδώ δηλαδή εμπεριέχεται η ουσία των όσων προσπαθούμε να κάνουμε, πάντοτε όμως συνεργαζόμενοι με τα ε, μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, πρακτική εφαρμογή των κεντρικών χρηματοδοτικών εργαλείων από τους NPBs να πούμε ότι έχουμε εμπλακεί ευθύ εξ αρχής στην, στο σχέδιο Juncker συνεργαστήκαμε δηλαδή με τους ε, φορείς ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Επενδύσεων ε, προκειμένου να βελτιώσουμε τις λεπτομέρειες και γενικότερα να ευθυγραμμίσουμε τα, τις υφιστάμενες πλατφόρμες και τα υφιστάμενα προγράμματα, τις δυνατότητες που δίνουν και τα τρέχοντα επενδυτικά σχέδια. Επίσης αναφέρουμε εδώ στην παρουσίαση μία σειρά από περαιτέρω εργαλεία, για παράδειγμα είχαμε ε, το Innov Fines που υπογράφηκε τον Μάιο του 2015. Επίσης ο NPP της Γερμανίας τον Ιούλιο του 2015 ε, υπέγραψε με συμφωνία ε, με το, για το κόσμο LGF οι, Πολωνίοι Πολωνοί συνάδελφοι ε, το 2015 επίση υπέγραψαν μια συμφωνία για αντεγγυήσει, πάντω στο επίθετο του κόσμου και αν θυμάμαι καλά, οι συνάδελφοι από την ε, Τσεχία ε, επίση προέβησαν σε μια συμφωνία για επενδύσει, για, για για ένα πρόγραμμα αντεγγυήσεων. Αυτά λοιπόν ω προ τα όσα κάνουν τα χρηματοδοτικά μέσα. Να πούμε τώρα, από τη δική μα πλευρά, εμεί τι κάνουμε. Έχουμε συμμετάσχει στι ε, διάφορες διαδικασίε εργασιών που έχουν δημιουργηθεί από την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε ό,τι αφορά δηλαδή εγγυήσει, αμοιβαία κεφάλαια, συμβουλευτικέ υπηρεσίε και ούτω καθεξής. Συμμετείχαμε και στις ομιλίε που έγιναν για την εκπόνηση του κανονισμού ε, για τα ΕΦΣΙ, τα Διαφθορτικά και επενδυτικά ταμεία και Ε, συνολικά 700 εκατομμύρια ευρώ καταφέραμε να εξασφαλίσουμε είτε μόνοι μας είτε μέσω ε, ε, σε συνεργασία με το Ταμείο Επενδύσεων. Και τώρα θα επισέλθω σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τα, τα προγράμματα εγγύσεων μας, ούτως ώστε να σας δείξω πού τα χρηματοδοτικά μας μέσα εξασφαλίζουν την προστιθάμενη αξία για χρηματοδότηση δηλαδή προγραμμάτων τα οποία ήδη υπήρχαν σε εθνικό επίπεδο. Ε, ε, η συμφωνία μας, η αυτό το πρόγραμμα ήταν το πρώτο που υιοθετήθηκε από το Ταμείο Επενδύσεων ε, στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker τον Μάιο του 2015 και υποστηρίζεται από το SME Window όπως λέγεται, δηλαδή το τμήμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του σχεδίου Juncker και αποτελείται από ένα χαρτοφυλάκιο 420 εκατομμυρίων ευρώ ε, ως δάνεια για καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ε, μικρά και μισά κεφάλαια. Έχουμε δύο τμήματα εδώ. Έχουμε καταρχήν το ε, δάνειο καινοτομία, το οποίο στοχεύει στο να προωθήσει τις καινοτομίες. Καινοτομίες δηλαδή από επιχειρήσεις οι οποίες είχαν ε, λάβει την υποστήριξη από προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Θεωρήσαμε δηλαδή ότι καλό θα είναι στα πρώτα στάδια ακριβώς της καινοτομία αυτές οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν υποστήριξη. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι το Seed Investment Loan όπως λέγεται, δηλαδή επενδύσεις σε κεφάλαιο εκκίνησης, το οποίο ε, ουσιαστικά συντονίζει την ε, εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων από ιδιώτες επενδυτές. Πώς τώρα αυτά τα δύο ε, προγράμματα εντάσσονται, αν θέλετε, στον γενικό μας προγραμματισμό. Εδώ, σε αυτήν τη ε, διαφάνεια, βλέπετε ποια ήταν τα προγράμματα μας πριν. Στα αριστερά, δηλαδή, βλέπετε τις ε, πρώτες φάσεις, δηλαδή την διατύπωση, την αξιολόγηση της το, το feasibility και ούτω καθεξής και στα δεξιά βλέπετε από εκεί και μετά τις, τις φάσεις της ανάπτυξης Είχαμε για παράδειγμα εδώ ε, δάνεια ανάπτυξης ε, τα οποία δόθηκαν από κοινού με εμπορικές τράπεζες. Στη μέση της διαφάνειας ε, βλέπετε έχουμε ένα κενό εδώ, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την γκάμα των χρηματοδοτικών προϊόντων που προτείνουμε και έτσι ακριβώς με τα, τα, τα, δύο νέα προγράμματα, δηλαδή τα ε, δάνεια καινοτομία και τα δάνεια κεφαλαίου εκκίνησης, γεφυρώνουν, αν θέλετε, αυτό το, το, το χάσμα μεταξύ των, ε, της χρηματοδότησης έρευνας και ανάπτυξης αφενός και των ε, δανείων ανάπτυξης αφενός, γιατί, ε, αφετέρου, γιατί τα δάνεια ανάπτυξης βέβαια είναι, έχουν αρκετά υψηλή επικινδυνότητα και κατά συνέπεια δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως το, το χάσμα χρηματοδότησης, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις νέες επιχειρήσεις. Ε, τώρα, ε, το feedback που έχουμε λάβει για αυτά τα προγράμματα ε, είναι, έχει υπάρξει αρκετά θετικό γιατί μόνο μετά από 9 μήνες έχουμε ήδη διαθέσει το 62% του, του χαρτοφυλακίου μας και έχουμε ήδη υποστηρίξει περισσότερες από 700 καινοτόμες επιχειρήσεις και έχουμε ήδη υποβάλει αίτηση για περαιτέρω χαρτοφυλάκιο. Τώρα, κλείνω την παρουσίασή μου με μια επισκόπηση των ε, χρηματοδοτικών μέσων με τα οποία εργαζόμαστε αυτή την περίοδο. Άρα λοιπόν πέρα από ε, το φίν, δηλαδή την, ε, το χρηματοδοτικό μέσο για τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Έχουμε εγγυήσεις οι οποίες δίνονται στον πολιτισμικό τομέα. Μετά έχουμε ε, τις εγγυήσει για μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις με πάνω από 500, 500 εργαζόμενους. Επίσης έχουμε ε, τις, ε, τα δάνεια για την χρηματοδότηση σε βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε mid-caps πάλι. Επίσης υποστηρίζουμε την ε, νέα ε, πλατφόρμα ENSI ε, για το, η πρωτοβουλία δηλαδή securitization του Ταμείου Επενδύσεων και των, των Εθνικών Τραπεζών Προώθησης. Επίσης έχουμε ένα νέο ε, ταμείο SPI όπως ονομάζεται ε, στην ε, Γαλλία και είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων για τις επενδύσεις στο μέλλον. Επίσης έχουμε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα τώρα για equity, για συμμετοχικά δάνεια. Και μία σειρά από προγράμματα εδώ και στον τομέα του δοχικού κεφαλαίου που σας δείχνουν ποιο είναι το χαρτοφυλάκιο το οποίο εμείς έχουμε ε, με τη μορφή των χρηματοδοτικών δηλαδή μέσων που μπορούμε να προσφέρουμε. Αυτά από την πλευρά μου και είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Μια σου λέγω μόνο. Αυτές οι κινήσεις και συναλλαγές που είπατε είναι εδώ να γίνουν χωρίς τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα, δηλαδή αν δεν υπήρχαν αυτές οι εγγύσεις, αν δεν υπήρχε η ευρωπαϊκή εγγύηση, τότε αυτά τα, τα, τα οποία κάνατε θα γινόντουσαν ή όχι. Ε, είναι δύσκολο το ερώτημα, λέει ο ε, καλεσμένος. Αυτό το πρόγραμμα ε, της προ δεν προβλέπεται, δηλαδή ε, είπαμε να το κάνουμε και είπαμε ότι θα έχουμε την πρικοδότηση και το μηχανισμό τον εγγυητικό που να είναι αρκετά στεγανός. Και ήταν και τότε που το κάναμε. Δηλαδή είπαμε τότε να υπάρξει μία προσφορά ε, όσο γίνεται πιο καλή για να καλύψει τις επιχείρησεις. Τώρα όσον αφορά τις ε, συναργίες μας που αφορούν το εταιρικό κεφάλαιο ή το μετοχικό κεφάλαιο, πριν αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ε, ε, ε, χρηματοδότησης είχαμε ένα παρόμοιο πρόγραμμα χρηματοδότησης με ένα πρόγραμμα για να καλυφθούν οι κοινοί στόχοι. Και έγινε μια αξιολόγηση ποσοτική για τις επιπλέον προστάσεις που να γίνουν για αυτό το πρόγραμμα το επενδυτικό για την Ευρώπη και κάναμε πολύ περισσότερα από όσα περιμένουμε. Τρεις φορές περισσότερο από την προστιθέμενη αξία είναι το ότι γίνανε περισσότερα και όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των εργαλείων, αυτή η προστιθέμενη αξία των νέων εργαλείων είχε εγγενή προστιθέμενη αξία. Είναι περίπλοκο. Και τώρα. Ο κ. Νομινίδη θα έχει το λόγο, είναι ο Γενικό Γραμματέα ε, του φορέα για ε, του ε, μακρόπνου επενδυτέ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να λάβω το λόγο ενώπιον σα, Η Ένωση Επενδυτών μακρά διάρκεια είναι στη φάση αναθεώρησης της διακυβέρνησής της, τώρα τα μέλη της, το Διευθυντικό Συμβούλιο θα παρτίζεται από τις Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες. Αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο είναι πολύ κατάλληλο για μια τέτοια ενέργεια. Θέλω να σταθώ στο ρόλο του φορέα μας και μετά θα θέσω τέσσερις ερωτήσεις επί τάπητος και θα σας αφήσω τρία μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, όταν μιλάμε για τις Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες και τα ιδρύματα αυτού του είδους, Προ το παρόν δεν υπάρχει ενιαίο ορισμό. δεν υπάρχει πραγματικός ορισμός. Μπορείτε να μου δώσετε αυτή τη διαφάνεια. Δεν υπάρχει, όπως είπα, ένας ενιαίος ορισμός του τι αποτελεί μια Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μπορώ να σας δώσω μονάχα μερικά γενικά στοιχεία που δεν είναι κατά ανάγκη ε, στοιχεία που να δείχνουν ότι όλες αυτές οι τράπεζες έχουν το ίδιο επιχειρηματικό μοντέλο, αλλά έχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα είναι δημόσιοι οργανισμοί με δημόσιο έλεγχο, αλλά συγχρόνως λειτουργούν σε εμπορική βάση και ακολουθούν τις ε, υγιείς τραπεζικές αρχές. Αυτό τις κάνει ε, σε σχέση με άλλους ε, διαμεσολαβητές στο χρηματοπιστωτικό χώρο. Ο στόχος τους δεν είναι η κερδοφορία, αλλά προώθηση των πολιτικών του δημοσίου και προφανώς γνωρίζετε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ πολιτικών και πολιτικής με μικρό πι. Εδώ οι τράπεζες αυτές θα πρέπει να είναι πολιτικά ανεξάρτητες ή θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητες και αυτό θέτει το ζήτημα της επιλογής των σχεδιών που χρηματοδοτούν. Σε εθνικό επίπεδο παίζουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχουν στόχο να ανταγωνίζονται τις άλλες εμπορικές τράπεζες στην αγορά, αλλά να αντιμετωπίσουν τις λεγόμενες αστοχίες της αγοράς και έχουν ένα, ε, μπορούν να έχουν ένα ρόλο ο οποίος είναι αντικυκλικός. Δύο βασικά στοιχεία της προστέμενης αξίας τους είναι το ότι έχουν μια ιδιαίτερη ικανότητα να αξιολογήσουν την αξία των επενδύσεων για το κοινό καλό. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την εμπορική προσέγγιση που είναι η οικονομική απόδοση μιας επενδύσεως. Εδώ μιλάμε για την προστιθέμενη αξία σε δημόσιο επίπεδο μιας επένδυσης και αυτό είναι βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση από τις τράπεζες αυτές και δεύτερον παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην παροχή συμβουλών λόγω της εμπειρίας τους και λόγω ορισμένων χαρακτηριστικών στα οποία θα επανέλθω μπορούν να φέρουν στην αγορά και συνεργασόμενοι και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορούν να δώσουμε συμβουλές για το καλύτερο τρόπο διάρθρωσης και χρηματοδότησης των σχεδίων. Δεν έχουν όλες το ίδιο επιχειρησιακό ε, μοντέλο, αλλά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα μακρόπνοα σχέδια επενδύσεων. Εδώ βλέπετε στην εικόνα αυτή την γέφυρα και είναι ακριβώς μια γέφυρα μεταξύ της κουλτούρας των δημόσιου τομέα και συγχρόνως των χρηματοδοτικών εργαλείων και της κουλτούρας της ιδιωτικής αγοράς. Πάνω από 30 χρόνια εργάζομαι στον τομέα αυτό και ξέρω ότι είναι μεγάλη η πολιτιστική διαφορά και χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να γεφυρώσουμε αυτές τις δύο κουλτούρες. Επίσης, έχουν πολλές φορές την ε, ε, καλύτερη γνώση για τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των τοπικών εταίρων και αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούν να συλλέξουν αυτή την πληροφορία πάντα. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να φέρουν πιο γρήγορα στην αγορά ορισμένα εργαλεία. Δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα τις 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την εξέλιξη του Λουξεμβούργου. Αυτό μπορεί να γίνει μονάχα με το να έχουν τοπική παρουσία. <clears throat> Τα περισσότερα κάτι μέλη έχουν μια Εθνική Τράπεζα ανάπτυξη και Επενδύσεων μέχρι τώρα σε ορισμένε περιπτώσει τώρα δημιουργείται μια τέτοια τράπεζα, είναι λίγε περιπτώσει που δεν υπάρχει. Με την παροχή λοιπόν βοήθειας από τις ε, ε, εθνικές τράπεζες ε, ανάπτυξης πράγματι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο όπως και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την εφαρμογή αυτών των σχεδίων. Έχουν πολλή εμπειρία Κάποιες από αυτές έχουν εμπειρία πάνω από 20 χρόνια για την εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων. Δεν θα σας αναφέρω όλα αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα από την αρχή, αλλά είναι σημαντική η εμπειρία που έχει σε αυτές τις ε, τράπεζες. Θα ήθελα τώρα να σταθώ στο ΕΦΣΥ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το οποίο δεν είναι απορριθμιστική έποψη χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά παίζει το ρόλο ενός χρηματοδοτικού εργαλείου. Δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση των ε, Εθνικών Αναπτυξιακών Τράπεζων στα, στις εγγύησεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Μέχρι στιγμή υπάρχουν τρεις δυνατότητες συνεργασία με το ΕΦΣΥ. Καταρχήν, συγχρηματοδότηση μεγάλων σχεδίων. Αυτό δεν αφορά όμως συνήθως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, η διαμεσολάβηση μεταξύ Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζες Επενδύσεων και Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και Μικρομεσαίων Επιχείρησεων. Και τρίτος τομέας, που για μένα είναι ακόμα κάπω ασαφής, <clears throat> είναι η δυνατότητα να εργαστούν μέσω πλατφορμών. Για μένα οι πλατφόρμες είναι αυτή τη στιγμή περισσότερο σύνθημα παρά πραγματικότητα. Υπάρχει πάντως η δυνατότητα να δημιουργηθούν πλατφόρμες όπου σε περιφερειακό επίπεδο ή σε επίπεδο τομέων αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης μπορούν να συμβάλλουν και θα συμβάλλουν στην παροχή πληροφοριών και συμβουλών μέσω του κέντρου ή του δικτύου παροχής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα τέσσερα ερωτήματα τώρα που θέλω να θέσω. Πρώτο ερώτημα είναι το εξή: Γιατί να χρησιμοποιήσουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποστηρίξουμε με εγγύηση στο ΕΦΣΥ και όχι τα διαφορετικά ταμεία ή τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Δεν θέλω να τονίσω ότι δεν χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής τα διαφορετικά ταμεία για να υποστηρίξουν χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά είναι απαραίτητο όπως έχει λεχθεί να απλοποιήσουμε τους κανόνες. Είναι απαραίτητη προτεραιότητα λοιπόν η απλοποίηση των κανόνων. <clears throat> Γιατί πολλά ιδρύματα, πολλοί παίκτες στην αγορά δεν χρησιμοποιούν τα χρηματοδοτικά αυτά γιατί είναι πολύ πολύπλοκα και πολύ, πολύ δάπανα στην εφαρμογή τους. Με μία διαφάνεια και μόνο. Το υπόδειγμα του FC <coughs> στα αριστερά έχουμε την πρώτη απώλεια στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά ε, το επόμενο επίπεδο απώλειας είναι στο Ευρωπαϊκό, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μετά είναι ο ιδιωτικό τομέα. Αυτό μπορεί να γίνει όμως και με τις Εθνικές Τράπεζες Ανάπτυξης να παίζουν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα μπορούσε να γίνει λοιπόν σε εθνικό επίπεδο. Γιατί, πώς λοιπόν θα εξασφαλίσουμε την προσθετικότητα και θα αποφύγουμε να βγάζουμε από το παιχνίδι τον ιδιωτικό τομέα. Βέβαια εδώ έχουμε τις επιτροπές του ΕΦΣΙ οι οποίες προσπαθούν να το αποφύγουν αυτό αλλά κάνουν κυρίως εστιάζουν περισσότερο στις ειδικέ δραστηριότητες με μεγάλο κίνδυνο όπως ε, αναφέρονται αυτές οι δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ο στόχος δεν είναι να αυξηθεί το σύνολο της δανειοδότησης γιατί αυτό το οποίο ενδιαφέρει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι το συνολικό επίπεδο επενδύσεων και όχι το συνολικό επίπεδο δανειοδότηση. Για τι εθνικέ αναπτυξιακέ τράπεζε παραμένει <clears throat> σημαντικό να μπορέσουν να βρουν το ρόλο του μέσα σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να μην υποκαταστήσουν τον ιδιωτικό τομέα. Ακόμα και όταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, παίζει το ρόλο ενός εταίρου που έχει πρώτη ε, δυνατότητα απώλειας και οι εθνικές τράπεζες σε δεύτερο επίπεδο, σε, πιο, σε επίπεδο πιο εξασφαλισμένο, πάλι αυτές οι τράπεζες παίρνουν το, τη θέση των ε, ε, ιδιωτικών φορέων. Θα έπρεπε να υπάρχει μια δυνατότητα εγγύησης των ε, εθνικών αυτών αναπτυξιακών τραπεζών που να έχουν ανάλογο ρόλο με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το τρίτο με ερώτημα τώρα είναι πώς θα εξασφαλίσουμε ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία πράγματι φτάνουν τα κράτη-μέλη και τους πελάτες που χρειάζονται περισσότερο αυτά τα δάνεια και όχι τους άλλους. <clears throat> και αυτό είναι ένα γνωστό θέμα. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει το ζήτημα του πολιτικού κινδύνου που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν έχω συναντήσει ούτε ένα θεσμικό επενδυτή που παρουσιάζει το θέμα αυτό ως το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όταν τους ζητούν να επενδύσουν σε ορισμένε χώρες, ότι υπάρχει πολιτικός κίνδυνος. Για να μπορέσει να ξεπεραστεί και αυτό το ερώτημα, αυτό το πρόβλημα, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ενίσχυση του ρόλου των εθνικών τραπεζών ανάπτυξης, γιατί αυτοί έχουν καλύτερη πρόσβαση στις απομεμακρυσμένες περιοχές και επιχείρησεις. Το τέταρτο ερώτημα μου είναι, πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε τις μικρότερες επιχειρήσεις και δυστυχώς αυτό είναι δύσκολο. <clears throat> Είναι σχεδόν αδύνατο να διαβάσετε τα αριθμητικά στοιχεία σε αυτήν τη διαφάνεια, αλλά θέλω απλώς να επιστήσω την προσοχή σας στα στοιχεία. 92,2% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικροεπιχείρησεις. 29,6% της απασχόλησης και 21% του ΑΕΠ είναι μικροεπιχείρησης. Ας μην ξεχάσουμε λοιπόν ότι υπάρχουν μικροεπιχείρησεις. Είδα ότι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μικροχρηματοδότηση ούτε καν αναφέρεται. Και υπάρχουν βέβαια κενά στη χρηματοδότηση. Είναι κρίμα που δεν δίνονται περισσότεροι πόροι για τις μικρές επιχειρήσεις. Υπάρχει και μια νέα πλατφόρμα για μετοχικό κεφάλαιο για τις μικρές επιχειρήσεις με το όνομα του Ελένος, που θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Ποια είναι τα συμπεράσματά μου σε τρία σημεία και μόνο. <clears throat> Πρώτα απ' όλα, και αυτό έχει αναφερθεί ήδη από την Πολωνίδα συναδελφό μου της BGK, οι χορηγήσει και τα χρηματοδοτικά εργαλεία πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Οποιαδήποτε προσέγγιση η οποία δεν διαφοροποιεί μεταξύ των δύο θα αποτύχει. Μπορεί κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία να έχουν και ένα στοιχείο ε, χορήγησης, αλλά γενικά έχουν διαφορετικούς κανόνες, διαφορετική επιλεξιμότητα και είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη την απαραίτητη αναλογικότητα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την παροχή αναφορών. Μόνο λοιπόν σε σχέση με το μέγεθος της χορήγησης και όχι της συνολικής χρηματοδότησης πρέπει να λάβατε αυτό υπόψη. Επίσης ένα άλλο παράδειγμα είναι το εξή Γιατί, γιατί έγινε και γίνεται ακόμα αυτή η τεράστια μάχη για την επαναχρησιμοποίηση των κονδυλίων όταν δεν λέει κανείς για την επαναχρησιμοποίηση των κονδυλίων μετά από μία χορήγηση. Δεύτερο μήνυμά μου είναι απλοποίηση και ευελιξία. Απλώς επαναλαμβάνω αυτά που είπανε και οι άλλοι ομιλητές, αλλά υπάρχει ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός εργαλείων και αναρωτιέται κανείς αν επικαλύπτονται αυτά και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να επιτύχουν την κρίσιμη μάσα που απαιτείται για να προχωρήσει αυτό το είδος και αν δεν μπορούν έτσι να χρησιμοποιήσουν τις δυνητικές συνέργειες. Τόσοι πολλοί εμπλέκονται. Η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο ανάπτυξη, οι εθνικέ αναπτυξιακέ τράπεζε, οι δικαιούχοι κτλ. Γενικά υπάρχουν διαφορετικέ νομικέ βάσει και διαφορετικοί κανόνε. Υπάρχει πολύ μεγάλο κίνδυνος να μπλοκάρονται τα πράγματα μόνο και μόνο λόγω τη σύγκρουση μεταξύ των κανόνων αυτών, ακόμα και όταν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, το κόστος για τις διαδικασίες, το κόστος για τις παρουσία πολλών εταίρων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Επομένως για τον επόμενο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε μια απλοποίηση του πλαισίου για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί δεν το βλέπετε από την οπτική γωνία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αυτό που θα οδηγήσει σε μεγάλη απλοποίηση. Και το τρίτο μήνυμα είναι βέβαια χρησιμοποιήστε καλύτερα τις Εθνικές Τράπεζες Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τους λόγους που θέλησα να <clears throat> εξηγήσω, γιατί βοηθούν σε μια προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω και έτσι συμπληρώνουν την εκ των άνω προς τα κάτω δράση των φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει και μια συνέχεια στα εργαλεία και στους κανόνες, γιατί υπάρχει και ένα κόστος επενδύσεων για αυτούς τους φορείς, όταν αρχίσουν να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία και πρέπει να τα αποσβέσουν εν καιρό και θα θέλανε να έχουν και ήδη και ίση μεταχείριση όλων, μεταξύ όλων των εμπίστων, όπως λέμε, φορέων. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τιακού. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Οπότε τώρα θα σας υποβληθούν οι ερωτήσεις από τους συναδέλφους που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις. Η κυρία Ρίεντα. Ήταν άρεστη η παρουσίαση και μας τα είπατε πάρα πολύ καλά. Μια ρωτησούλα. Μας λέτε για τις πολιτικές των Εθνικών Τραπεζών πρόθεση. Ποιος χαράσε αυτές τις πολιτικές. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει αποστασιοποίηση από την πολιτική. Αλλά ξέρουμε πολλές φορές που λειτουργεί το σύστημα. Εσείς συμφωνείτε ότι πρέπει έτσι να γίνεται. Άλλες ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Επομένως, το μήνυμά σας επικεντρώνεται το ότι χρειάζεται απλούστευση. Όσο γίνεται περισσότεροι ε, απλούστευση αλλά και σταθερότητα στις ρυθμίσεις που είναι η μόνη σύνταχη ούτως ώστε ε, είναι κατανοητό το πλαίσιο και έτσι να βοηθούνται οι επενδύσεις για τέτοιου είδους ε, μακροπρόθεσμη δανειοδότηση. Όμως, από όσο μας είπατε φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο. για τις συναλλαγές σε ευρωπαϊκό ε, να μπορούν άμεσα να εισπράξουν ε, ε, αυτόν τον δανεισμό οι ΜΜΕ, γιατί υπάρχουν οι τράπεζες οι οποίες είναι διάμεσες και οι οποίες αναβαίνουν τον κίνδυνο. <coughs> Παρ' όλα αυτά, πιστεύετε ότι έχουμε τάση κινητοποίησης ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα το επενδυτικό από το οποίο υποφέρει η Ευρώπη εδώ και 10 χρόνια ή παραπάνω, με τα μέσα που έχετε στη διάθεσή σα μπορείτε να επιταχύνετε τι ε, εξελίξεις, να το πάρετε ούτως υπήρει την κατάσταση. Βέβαια για τι τράπεζε είναι πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Έτσι δίνονται εγγύησεις, συναπτώνται δάνεια από τη βάση των εγγύσεων και όσον αφορά τις κρατικέ επενδύσεις είναι δυνατόν να προχωρήσουν όπως και το δημοσιο χρέος. Βέβαια υπάρχουν και κίνδυνα που μας είπατε κύριε Κρένκουλ, Υπάρχει ε, αυτό το, το, το πρόβλημα της εμπιστοσύνης. Αλλά ο κερδισμένος είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κερδισμένο, αλλά με την καλή έννοια. Δεν βλέπω να ζητεί άλλο το λόγο. Οπότε, αν θέλετε, να διευκρινίζετε αυτά που εξήγησατε. Ναι, ναι, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι μέλος της ε, Επιτροπή για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και αυτή την περίοδο ε, ετοιμάζουμε μία έκθεση ε, εφαρμογής και ένα πολύ σημαντικό τμήμα αυτής της έκθεσης αφορά την εφαρμογή ακριβώς των χρηματοδοτικών μέσων. Γι' αυτό και θεώρησα αυτή την εδώ και την όλη συζήτηση που έγινε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για τη δουλειά που κάνω εκεί στην Επιτροπή δηλαδή. Και βέβαια για το έργο που κάνει η, Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό της. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και πάντοτε τα συμπεράσματα είναι ίδια. Δηλαδή ότι δεν είναι αρκετά στοχευμένο ο κανονισμό, δεν υπάρχουν αρκετέ εξηγήσει, δεν υπάρχει τυποποίηση, συνέχεια ε, γίνονται τροποποιήσει και ούτω καθεξή. Αλλά θα ήθελα να ακούσω από εσά περισσότερα. Ε, Εσεί προέρχεστε από το τομέα τη πρακτική εφαρμογή, αν θέλετε. Άρα, ε, ποια είναι τα πρακτικά εμπόδια που αντιμετωπίζετε. είναι για παράδειγμα οι κανόνε κρατικών ενισχύσεων που δημιουργούν τέτοιου είδου προβλήματα. Γιατί ξέρω, για παράδειγμα, ότι στη δική μου χώρα, στην Κροατία, όταν δίνονται ενισχύσει για καινοτομία και η ε, λαμβάνονται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από δημόσιες αρχές για την καινοτομία. Ε, η χρηματοδότηση λαμβάνεται ε, κατά 50% αλλά το υπόλοιπο 50% δεν μπορεί να ληφθεί μέσω χρηματοδοτικών μέσων γιατί θεωρείται και πάλι κρατική επιχορήγηση. Άρα τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί να γίνει δηλαδή ένα είδος ε, ε, δημόσιας σύμβασης μια αντίστοιχη διαδικασίας γιατί τελικά δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι τελικά η τυποποίηση. Δηλαδή, ε, σίγουρα πάντοτε χρειάζονται κάποιες εξειδικευμένες ε, διατάξεις για να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες, αλλά σε αυτό το επίπεδο που μου ανέφερα μόλις τώρα ενδεχομένως θα ήταν δυνατό, δηλαδή της πρακτικής εφαρμογής, να επιτύχουμε κάποια βελτίωση. Αυτό είναι μια ευχή που την να πούμε και τη συμμεριζόμαστε όλοι. Κάθε μέρα λέμε. Απλούστευση. Μια που είναι κολλημένη σε αυτή τη γραφειοκρατία, σε αυτή την πληθώρα των νομικών βάσεων η Ευρώπη και δεν μπορεί να λάβει τι ε, αποφάσει. Οπότε και η προσδοκόμενη ε, απάντηση είναι ότι πρέπει να σταματήσει υπάρχει αυτή η αδράνεια. Βέβαια δεν είναι άσχημα αυτό δημοσιονομικά, γιατί έτσι όπως είμαστε κολλημένοι, και δεν προχωράμε, δεν ξοδεύουμε χρήματα. Βέβαια, δεν είναι αυτό ο στόχος. Δεν θέλουμε να πάμε προς τα εκεί. Τώρα, η κύριε Ντιμπαρή και η κυρία Νικούρ, μήπως μπορείτε πάρα πολύ σύντομα να απαντήσετε σε αυτά τα οποία ερωτήθηκαν από την κυρία Ριάντα, από την συνάδελφο της Περιφερειακής Επιτροπής, και την ερώτηση του υποφαινομένου και κατόπιν θα συνεχίσουμε με το τελευταίο τμήμα της ε, συνάντησης. Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, εμείς παραβαίνουμε χρησιμοποιώντας αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο και υπάρχουν ε, διατάξεις ούτως ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερες επιχειρήσεις σε κλάδους και τομείς ιδιαίτερα πολλού κινδύνου. Και ε, παρεμβαίνουμε στην ε, αγορά επίσης στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι τόσο άσχημο το ρυθμιστικό πλαίσιο. Να συμμετάσχουμε, να το βελτιώσουμε. Τώρα θα σας τα πει και ο Ντομίνικα, αλλά όσον αφορά ε, τις την Ευρώπη, και το, ρόλο του ενδιαμέσου είναι δύσκολος ο ρόλος. Χρειάζεται απλούστευση αλλά και ένας άλλος στόχος σε αυτό το, το περιβάλλον, αυτό το οικοσύστημα είναι ε, η προσαρμογή στο, στις εθνικές Οπότε να υπάρχει μια συνέργεια μεταξύ των ε, εργαλείων των ευρωπαϊκών και των εθνικών και έτσι να ενεργοποιηθεί η μόχλευση και όλα μαζί να αποδίδουν. Αυτό είναι δύσκολο βέβαια γιατί αυτά τα εργαλεία ε, έχουν φτιαχτεί στην Ευρώπη οπότε δύσκολα να καλύψουν 28 διαφορετικές ε, ανάγκες αλλά στο επίπεδο της εφαρμογή ε, να υπάρχει ευελιξία και για να υπάρχει προσαρμογή σε κάθε χώρα. Σας είπα και τις προσπάθειες του ομίλου της ε, ΕΤΕ για να ανταποκριθούμε στο τι χρειάζεται κάθε χώρα σε σχέση με αυτά τα εργαλεία. Και από έχουμε το ε, γραφείο και των καταπιστευμάτων, το άλλη μεριά έχουμε το κράτος και δουλεύουμε με αυτά τα αφεντικά, συνεργαζόμαστε και με τα περιφερειακά συμβούλια όσον αφορά την προσφορά των υπηρεσιών για κάποιες ε, περιφέρειες που συμμετέχουν και αυτές στην διακυβέρνηση που κάνουμε. Συνεργασία επομένως είτε με Ευρωπαϊκή Αρχή, είτε Εθνική, είτε Περιφερειακή. Ναι, αλλά η Περιφέρεια πολλές φορές έχει τους δικούς τους κανόνες για την χορήγηση αυτών των ενισχύσεων. Όχι άλλη νομοθεσία, αλλά κάποια άλλα εργαλεία τα οποία θέλουν να εφαρμοστούν, να χρησιμοποιηθούν για τις τοπικές ανάγκες. Αν δεν γίνεται πιο απλούστερα τα πράγματα έτσι. Να σας ευχαριστήσω για το πρώτο ερώτημα του ποιος κυβερνά τις πολιτικές των Εθνικών Τραπεζών Ανάπτυξης σε γενικές γραμμές είναι η κυβέρνηση της χώρας τους που καθορίζει την αποστολή τους επί τη βάση των εθνικών πολιτικών. Προφανώς όμως όταν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι τα διαρθρωτικά ταμεία και έχουν κεντρική διαχείριση, εκεί επικρατεί η ευρωπαϊκή πολιτική και ελπίζω ότι δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση, κάτι το οποίο είναι σαφές, είναι ότι λόγω της αποστολής τους αυτοί οι φορείς δεν θέλουν ως, δεν θέτουν ως προτεραιότητα την κερδοφορία των οργανισμών τους. Αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ αυτών και των εμπορικών τραπεζών. Για το θέμα της, ε, του επίπεδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περισσότερο απάντηση ή παραρώτηση αυτό που δώσατε κύριε Πρόεδρε. Αλλά υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό. Και σκεφτείτε όλα τα επίπεδα που δεν εφαρμόζονται πάντα στι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν να κάνουν περισσότερο με τι υποδομέ. Σκεφτείτε την Ένωση Αγορών που έχει τεράστια επίπτωση και η Τραπεζική Ένωση βέβαια έχει επίπτωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε ακούσει για δράσεις που ξεκινούν από μια τράπεζα σε μια χώρα αλλά απευθύνονται σε άλλες χώρες. Ένα άλλο θέμα είναι η τίτλοποίηση. Αν δεν το έχετε σε επίπεδο της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον δεν αξίζει τον κόπο να, να μπείτε στον κόπο να το κάνετε. Και το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας είναι κατά πόσο με τον τρόπο αυτό δίνεται μία απάντηση στο αν αυτό είναι το πρόβλημα. Και ποιος είμαι εγώ να σας απαντήσω. Το πάνελ του σχεδίου Juncker δεν είναι μονάχα αυτός που δίνει τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Το πιο σημαντικό, ο πιο σημαντικός πυλώνας είναι και οι διαρθρωτικές αλλαγές, όλες οι άλλες πτυχές που θα κάνουν ευεπίφορο το, το πλαίσιο για τους επενδυτές να επενδύσουν. Αλλά μετά έχετε και τους κανόνες της Βασιλείας, τις απαιτήσει κεφαλαίου για τις τράπεζες. Αυτό οδήγησε σε απομόχλευση στις τράπεζες και έτσι άνοιξε αυτό το χάσμα στην αγορά και οι δύο λοιπόν πλευρές εδώ πέσουν και για τα προσκόμματα. Ο κύριος Ντιμπαρή απήντησε προηγουμένως. Δεν νομίζω ότι η λύση είναι πιο, ότι το πρόβλημα είναι πιο πολύ οι κρατικές επιδοτήσεις και οι κανόνες που τις συνοδεύουν, το σύνολο των κανόνων. Εγώ κοίταξα προσεκτικά το έγγραφο κατεύθυνσης που δόθηκε για το πώς να συνδυάζει κανείς τα διευθυντικά ταμεία με το ΕΦΣΥΧ. Χρειάστηκα σπυρίνες προτού να φτάσω στο τέλος και δεν μπορούσα να διαβάσω όλο αυτό το κείμενο. Λείπαμε πάρα πολύ και μεταξύ των μελών μας. Έχουμε τέσσερα ή πέντε ή έξι μεγάλα ιδρύματα που έχουν αρκετό προσωπικό με, για ανθρώπους που έχουν το χρόνο και τη δυνατότητα να τα διαβάσουν όλα αυτά. Αλλά σε χώρες με μικρότερους φορείς δεν μπορούν να κάθονται να τα διαβάσουν. Είναι μια πλήρης επένδυση χρόνου για να το κάνω αυτό. Να πάω τώρα στην άλλη άκρη. Η μικροχρηματοδότηση, την οποία ανέφερα προηγουμένω κανονικά, ένα ίδρυμα μικροχρηματοδοτούμενο, έχει μεταξύ, 10, ε, μεταξύ 5 και 15 άτομα και του ζητούν να υπογράψουν μια σύμβαση με ένα φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οποίο χρειάζεται να βρουν ένα δικηγόρο. Συνήθω δεν έχουν πια ούτε καν ένα δικηγόρο ο οποίο να μπορέσει να διαβάσει ένα τόσο ογκώδε έγγραφο για να κάνουν μια συμφωνία. Προτιμούν να μην κάνουν τίποτα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά του κοστίζει πάρα πολύ να το κάνουν. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση επομένως δημιουργεί θέσεις απασχόλησης με τον τρόπο αυτό γιατί πολλαπλασιάζει τις θέσεις των εμπειρογνωμόνων για να ετοιμάζουν τους φακέλους και να ανταποκρίνονται στις ε, θελήσεις της Κομισιόν. Αυτό είναι μια άποψη που μπορεί να την υποστηρίξει και το Κοινοβούλιο. Υπάρχει μια ιστερία αριθμιστικού χαρακτήρα. Ο καθένας θέλει να μπορεί να πει ότι τήρησε τους κανόνες ακόμα και αν το τελικό αποτέλεσμα είναι καταστροφικό. Αυτή την κουλτούρα ίσως πρέπει να αλλάξουμε. Θα πρέπει να κλείσουμε τώρα και τη δεύτερη φάση και να περάσουμε στην τελική συζήτηση που θα έχουμε δύο παρεμβάσεις 10 λεπτών η καθεμία και όχι παραπάνω γιατί έχουμε καθυστερήσει. Ο πρώτος ομιλητής ο κύριος Σίμους που τον ακούσαμε προηγουμένως ο οποίος είναι εμπειρογνώμων για την ανταγωνιστικότητα από το Banking Forum της Ιρλανδίας και είναι ο ιδρυτής της Διεθνούς Συμμαχίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και μετά το Ρεμί Σαριέ, ο οποίος θα λάβει το λόγο εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Τραπέζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Κύριε Μάιερ, έχετε το λόγο. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μας δίνετε την uh, δυνατότητα να πούμε και εμεί δύο λόγια από την πλευρά μας. Ε, ήταν, ε, υπήρξε ένα ενδιαφέρον απόγευμα ε, και βέβαια εγώ μπορώ να αναφερθώ πολύ περισσότερο στην Ιλανδία από ότι σε οποιαδήποτε άλλο κράτο ε, μέλος ε, ε, σε ό,τι αφορά το τραπεζικό τομέα και βλέπουμε ότι έχουν, πραγματικά δεν έχει δοθεί κατάλληλη προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλη αυτή η χρηματοδότηση και τα μέσα που προβλέπονται για τη διευκόλυνσή τη είναι πολύ ενθαρρυντικά και ε, δεν μπορώ πραγματικά να αδικήσω τα όσα υπόθηκαν σήμερα σε σχέση με αυτό το ζήτημα, αλλά σε ό,τι αφορά ειδικότερα την ε, περίπτωση της Ιρλανδίας και ε, το ζήτημα της περαιτέρω ανάπτυξης των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων τους, πραγματικά έχουμε μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή, για να δούμε ποια είναι η οικονομική κατάσταση. Αν δούμε τις άμεσες ξένες επενδύσεις, ε, και πολλοί βέβαια λένε ότι εδώ είμαστε ένας φορολογικό παράδεισο για διεθνείς επιχειρήσεις, ε, αλλά δεν θα το συζητήσουμε. Εάν λοιπόν ναι, ότι το λένε πολλοί ότι πραγματικά αποτελεί φορολογικό παράδεισο η Ιρλανδία για τις ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ναι, ε, περιπτώσει Ε, αυτό ε, προσπαθούσα να πω είναι ότι εάν δεν λάβουμε υπόψη μα τι άμεσε ξένε επενδύσει, τότε η, Ιρλανδία, η κατάσταση, οικονομική κατάσταση τη Ισλανδία είναι πάρα πολύ κακή. Και ε, η, καταστροφή δηλαδή του τραπεζικού τομέα ε, υπήρξε πολύ μεγαλύτερη από τι άλλε χώρε, όπω για παράδειγμα στη Γερμανία. Δηλαδή δεν έχουμε ε, κάποια ε, τραπεζική δραστηριότητα σε επίπεδο κοινοτήτων, community banking. Έχουμε κάποιε τραπεζικέ ενώσει, οι οποίε όμω είναι πολύ περιορισμένε, δεν μπορούν δηλαδή να δανειοδοτούν μικρομεσαίε επιχειρήσει, είναι περιορισμένα τα κονδύλια τα οποία μπορούν να επενδύσουν έω 200.000 ευρώ, δεν μπορούν να προβούν σε υποθήκε. Οπότε το πρόβλημα που δημιούργησε η κατάρρευση των τραπεζών της Ιρλανδίας και ο αντίκτυπος που είχε ε, στο ε, κοινωνικό-οικονομικό ιστό της χώρας μας δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Αυτό λοιπόν που, λέμε, που είπαμε, μάλλον είπαμε ότι πήραμε μόνο αυτόν τον πυλώνα των τραπεζών και είπαμε ότι θα πρέπει σε κάποια, κάθε περίπτωση να ε, ανακάμψει και τους επιτρέπουμε να χρεώνουν τα υψηλότερα επιτόκια σε ό,τι αφορά ε, δανειοδοτήσεις, υποθήκες και ό,τι καθεξής. Αλλά αυτό δεν είναι επικοδομητικό. Αυτό δεν υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μα ούτε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις μας. Ε, και βέβαια το δικό μας πρόβλημα της Ιλλανδίας, είμαστε μια πολύ μικρή χώρα. Δηλαδή, οι τράπεζες που έχουμε, αυτές οι λίγες τράπεζες που έχουμε, είναι πραγματικά πάρα πολύ παράξενο αυτό που κάνουν. Δηλαδή, αναγκάζουν πολλές, εκατοντάδες και χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κλείσουν ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι ε, περιφερειακές ε, οργανώσεις προσφέρουν περισσότερη χρηματοδότηση από άλλα ε, ταμεία κερδοσκοπικά. Άρα ε, το ερώτημα που τίθεται είναι τελικά τι γίνεται, γιατί κανένας δεν κάνει κάτι ενάντια σε αυτήν την τάση του να εξαφανίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, και ε, μία παγκόσμια οργάνωση ε, είπε για την Ιρλανδία ότι οι ζητήματα και ε, διαφθοράς μέσα στην, ε, στο τομέα της νομοθεσίας επηρέασαν τη δημιουργία του νομικού πλαισίου. και βέβαια μία σειρά από ζητήματα τέτοιας πολιτικής διαφθοράς επιτρέπουν στους αρμόδιους για τη χάραξη της πολιτικής να εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα από ότι το δημόσιο συμφέρον. Και αυτά είναι λοιπόν τα βασικά προβλήματα εδώ που αντιμετωπίζουμε στην Ιρλανδία και γι' αυτό έθεσα προηγουμένως τα ερωτήματα ερωτήματα σε ό,τι αφορά το Ελλανδικό ε, Ταμείο ε, Στρατηγικών Επενδύσεων και την, ε, τράπεζα, την Ένωση Τραπεζών Χρηματοδότησης. Γιατί αυτά τα κονδύλια, αυτά τα χρηματοδοτικά κονδύλια τελικά δεν κατευθύνονται εκεί που πρέπει. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για παράδειγμα, ο ένας από τους δύο φορείς που σας ανέφερα υπόκειται στην, στη διαχείριση της Bank of Ireland και από το ε, ε, επιστοτικό οργανισμό. Οπότε ε, είναι πολύ λίγοι εκείνοι οι οποίοι τελικά δεν έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα με τέτοιου είδου χρηματοδοτήσει και με αποτέλεσμα βέβαια να μην είναι δυνατόν να απευθυνθούν τώρα σε αυτόν τον φορέα αφού αυτό σε κάνει από τη διαχείριση τη Bank of Ireland. Το Ταμείο Στατιστικών Επενδύσεων με τη σειρά του λαμβάνει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για να τα σε, και ο σκοπός είναι να τα δυνατοδοτήσει σε τρίτους αλλά όταν η δανειοδότηση γίνεται με επιτόκια, ε, ε, με τόκους, ε, επιτόκια 12 13% πραγματικά θα καθιστά αδύνατο να τα, να τα Δηλαδή, το, κόστο, το, το κόστος βάσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το υψηλότερο στην Ιρλανδία από ό,τι στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Οπότε δεν μπορούν να καταβάλουν επιτόκια της τάξης του 15% και του 20%. Και ένα ακόμα ζήτημα για το οποίο πολύ συχνά δεν θέλουμε στην Ιρλανδία να γίνεται λόγο, είναι ε, να ε, επιτρέψουμε ακριβώ τη δημιουργία του community banking και είναι πολύ εντυπωσιακά τα όσα ακούσαμε από τη, ε, από τη Γερμανία, δηλαδή ότι το 70% τη οικονομία στη Γερμανία χρηματοδοτείται από το τραπεζικό τομέα του community banking, ενώ εμεί, στην Ιρλανδία το 90% τη χρηματοδότηση της οικονομίας γίνεται από δύο μεγάλε τρύπε, οι οποίες ακριβώ χαρακτηρίζονταν από αλαζονία και από κακή διαχείριση και οδηγήθηκαν τελικά στην κατάρρευσή του. Άρα λοιπόν με βάση τα όσα ακούσαμε εμεί εδώ σήμερα πρέπει να πούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας και ο σχετικοί κλάδοι στην, ε, στη δική μας χώρα δεν πρόκειται να ανθίσουν, δεν πρόκειται να αναπτυχθούν εάν δεν δημιουργήσουμε ε, community banking. Ε, και εδώ μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και οι τραπεζικές ενώσεις. Όμως γιατί οι κυβερνήσεις η μία μετά την άλλη περιορίζουν ε, όλο ένα και περισσότερο στι τραπεζικέ ενώσει. Γιατί δηλαδή εφαρμόζουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά ε, ε, στις, ε, σε αυτές τις Ε, δηλαδή στι τράπεζε και αφετέρου σε αυτέ τι ενώσει του community banking. Υπάρχουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν διατίθεται, δεν κατευθύνονται δηλαδή στην πραγματική οικονομία. Ακριβώ λόγω των περιορισμών που υπάρχουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξετάσει κάποιο τελικά την περίπτωση που κυριαρχεί ε, στην Ιλλανδία και να κάνει ό,τι μπορεί ούτω ώστε να επιτρέψουμε ε, την χρηματοδότηση με χαμηλά επιτόκια μέσω τέτοιου είδου ε, χρηματοδότηση από κοινότητα του community banking, γιατί αυτό θα βοηθήσει και τον αγροτικό τομέα τη Ιρλανδία και θα αποτελέσει ένα κεντρικό ε, βήμα για την ανάπτυξη της εγχώριας τραπεζικής αγοράς στην Ιρλανδία. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η πτυχή σε κάθε περίπτωση να ενσωματωθεί ε, στα όσα θα κάνουμε στο επίπεδο της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής. Οτιδήποτε κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ θετικό. Και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήματα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάιερ. Φαίνεται ότι το τραπεζικό σύστημα έχει δυσκολίες στο να δώσει τις πιστώσεις σε επιτόπιο επίπεδο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά μόνο σε επιτόκια τα οποία είναι απαγορευτικά, ενδεχομένως να αντισταθμίζουν κάποιο κίνδυνο, δεν ξέρω. Θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Ρένε Ρεμί ο οποίος θα μπορούσε ίσως τα λόγια του να μας πει πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό, ποιο είναι το εξόδες του συστήματος σε ορισμένες χώρες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να ευχαριστήσω και την ευκαιρία που δίνεται στην ομάδα μας να συμβάλλουμε σε αυτήν την ε, συνάντηση. Λέγομαι Ρεμί Σαριέ, δουλεύω για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων που είναι μια θηγατρική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το οποίο ε, εν μέρη είναι ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ομάδα μου έχει σαν στόχο να συζητήσει για τα χρηματοδοτικά εργαλεία στις περιοχές όπου εμείς είμαστε ένας από τους φορείς που συμμετέχει όπως το κόσμο και το Horizon 2020. Και επίσης το σχέδιο Juncker, το EFSI. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η σύνολη ομάδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι φορείς οι οποίοι εστιάζονται ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε ομάδες ερευνητικού χαρακτήρα οι οποίες ελέγχουν κάθε δύο, δύο φορές ε, το χρόνο ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση και τα πορίσματα αυτής της έρευνας είναι πάντα περίπου τα ίδια. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα γιατί όταν θέλουν να πάρουν χρηματοδότηση από τις τράπεζες ακόμα και αν το σχέδιο που παρουσιάζουν είναι θετικό αν δεν έχουν κάποια εγγυητικά στοιχεία ή κάποια εγγύηση από κάπου αλλού είναι πολύ δύσκολο να πάρουν κάποιο δάνειο. Σε επίπεδο μετοχικού κεφαλαίου ξέρουμε ότι είναι υποκεφαλαιοποιημένες οι μικρομεσαίες στην Ευρώπη όταν μιλάμε για το ε, κεφάλαιο σύμπραξης επιχειρήσεων, το οποίο συγκροτείται κάθε χρόνο στην Ευρώπη, είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια ε, ευρώ. Για το σύνολο της Ευρώπης, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 50 δισεκατομμύρια. Είναι πάνω από 10 φορές περισσότερο το αντίστοιχο κεφάλαιο που αφορά συμπράξη για την ανάληψη κινδύνου. Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα για τις μικρές επιχειρήσεις να πάρουν και είτε μετοχικό κεφάλαιο είτε δανειοδότηση από την πλευρά τη ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Εμεί δεν συνεργαζόμαστε άμεσα με τι ε, μικρομεσαίε παρά έμεσα. <clears throat> Λειτουργούμε μαζί με του εταίρου που είδατε προηγουμένω, δηλαδή τι Εθνικέ Τράπεζε Ανάπτυξη, τι Εμπορικέ Τράπεζε, του Φορεί Εγγυοδοσία και νομίζω ότι είναι πολύ καλή συνεργασία μα μαζί του. Χρειαζόμαστε αυτή τη συνεργασία για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζα, μάλλον Τράπεζας Επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση το 2015, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έδωσε 28 δισεκατομμύρια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καλύπτοντας περίπου 240.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που, που απασχολούν πάνω από 5 εκατομμύρια ανθρώπους σημαντικός αντίκτυπος για τα χρηματοδοτικά τώρα εργαλεία. Πρέπει να παραδεχτώ ότι τα εργαλεία αυτά προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εργάζονται πολύ καλά. Το πρόβλημα που έχουμε είναι η έλλειψη προϋπολογισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πληθώρα προϋπολογισμού και δυνατοτήτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το κόσμο. Το κόσμο αντιμετωπίζει πιο πολύ ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και είναι αυτές οι οποίες δυσκολεύονται πολύ να βρουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Το κόσμο βοηθάει να έχουν πρόσβαση στις τράπεζες. Το Ινοφιλ επίση είναι πολύ επιτυχές αυτό γιατί αφορά τις καινοτόμες επιχειρήσεις και πρέπει και οι τράπεζες να συμφωνήσουν ότι είναι καινοτόμα τα σχέδια που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις αυτές και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και στην πράξη αυτή τη στιγμή είναι 500 οι μικρομεσαίες οι οποίες έχουν πάρει κάποιο δάνειο που υποστηρίζεται από κάποιο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το ΕΦΣΙ, το σχέδιο Juncker, μετά από 9 μήνες που ξεκίνησε το σχέδιο αυτό, ε, το σχέδιο αυτό θα καλύψει 36 μήνες συνολικά. Η ομάδα της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων έχει εγκρίνει ε, διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε 82 δισεκατομμύρια ευρώ ή περίπου 26% του στόχου. Σε ό,τι αφορά το χρονικό διάστημα, σε 9 μήνες είμαστε περίπου στο 1 τέταρτο του συνόλου. Για τις μικρομεσαίες, για το παράθυρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μπορούμε να πούμε ότι θα εφαρμοστεί πλήρως ένα χρόνο πριν από την εκπνοή του. Σήμερα εγκρίναμε ε, ε, χορηγήσουμε με το παράθυρο της, ε, των μικρομεσαίων σε 26 χώρες. Μόνο την Μάλτα και την Κύπρο δεν έχουμε χρηματοδοτήσει αυτή τη στιγμή, αλλά θα καλυφθούν και αυτές η Ιλλανδία Η Τράπεζα της Ιλανδίας έχει υποστηριχθεί από αυτό το εργαλείο και μετά μπορεί να δώσει πρόσβαση σε χρηματοδότηση στις μικρομεσαίες επιχείρησης 137.000 δικαιούχοι θα είναι από την πλευρά των μικρομεσαίων και δεν έχουν τελειώσει όλα αυτά. Θα συνεχίσουμε την ανάπτυξη αυτού του προγράμματο και χάρη στην υποστήριξη τη Κομισιόν μπορούμε να αυξήσουμε επιπλέον την ικανότητα χωρί χρηματοδότησή μα. Έχουμε υπογράψει συμφωνίες εγγύηση με πάνω από 70 διαμεσολαβητικούς φορείς και επίσης και με περαιτέρω ιδιωτικά ταμεία. Οι χώρες οι οποίες έχουν τα κύρια θετικά αποτελέσματα είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία. Αλλά αν δείτε κατά κεφαλή, κυρίως η Σλοβενία, η Εστονία και το Λουξεμβούργο παίρνουν την περισσότερη κατά κεφαλή χρηματοδότηση. Υπάρχουν ακόμα πολλές ανάγκες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν, κυρίως στον τομέα του μετοχικού κεφαλαίου της μικροχρηματοδότησης μαζί με την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσπαθούμε να αναπτύξουμε και νέα εργαλεία μέσα στο ΕΦΣΥ ένα για, την, ε, το μετοχικό κεφάλαιο και ένα για τη μικροχρηματοδότηση και υπάρχουν και άλλα εργαλεία τα οποία θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην αγορά όπως αυτό για τον πολιτιστικό τομέα στις μικρομεσαίες επιχείρησεις. Από την πλευρά λοιπόν των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά. Σίγουρα τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα σε επίπεδο διαδικασίας. Θέλουμε πάντα κάθε τράπεζα να αναφέρει την, το ταχυδρομικό κώδικα της έδρας της ε, μικρομεσαίας επιχείρησης. Το χρειαζόμαστε αυτό πράγματι. Ναι, το χρειαζόμαστε στο λογιστικό έλεγχο να μπορέσει να φτάσει ω εκεί και να κάνει τον έλεγχο, αλλά οι τράπεζε σε όλε τι ε, δοσοληψίε του μα δίνουν αυτέ τι ε, πληροφορίε. Τα καλύτερα εργαλεία μας λοιπόν είναι αυτά όπου οι μικρομεσαίε μαζί με την Κομισιόν μπορούν να συναντηθούν και μαζί με τους ε, χρηματοπιστωτικούς ενδιάμεσους για να εντοπίσουν τα χάσματα που βρίσκονται στην αγορά και να βρουν τρόπους να υποστηρίξουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση της δημιουργικής Ευρώπης, της χρηματοδότησης πολιτιστικών φορέων, αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Ξεκινήσαμε με τις μικρομεσίες λέγοντας κάθε φορά που πάω στην τράπεζά μου, η τράπεζά μου μου λέει δεν καταλαβαίνω τι κάνετε εδώ πέρα, έχετε άειλα στοιχεία ενεργητικού, δεν ξέρω πώς να τα μετρήσω, δεν ξέρω ποια θα είναι η ταμιακή σας ροή που θα προκύψει από τα πνευματικά σας δικαιώματα. Μπορείτε να μου δώσετε λοιπόν το σπίτι σας ως ενέχειρο. Και επομένω αυτό ο τομέα βρίσκεται σε μεγάλη δυσκολία. Γιατί αυτέ οι μικρομεσαίε που είναι πολύ μικρέ συνήθω δεν έχουν πάντα ένα επιχειρηματία στη επικεφαλή που να έχει μεγάλη προσωπική περιουσία. Ακούγοντα αυτά που είδαμε σήμερα, είναι φανερό ότι υπάρχουν πολλές ε, διαφορές μεταξύ των χρηματοδοτικών εργαλείων με κεντρική διαχείριση και αυτών με επιμερισμένη διαχείριση. Στην περίπτωση επιμερισμένης διαχείρισης βασίζεται κανεί περισσότερο στα διαφορετικά ταμεία και εκείνη τα πράγματα πολύ πιο πολύπλοκα στην εφαρμογή τους έχουν σαν στόχο για χορήγηση και είναι και πολύ δύσκολο να, τις, να τους προσαρμόσουμε σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν είναι πρόσφορος λοιπόν ο κανονισμός για κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Και εν γέννη θα έλεγα ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι πολύ χρήσιμα. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για την χρήση αυτών των εργαλείων και σε τελική ανάλυση ένα ευρώ δημοσίου χρημάτων οδηγεί σε 10 ή 20 ευρώ ε, δανείων. Και αυτό οδηγεί σε απασχόληση και ανάπτυξη. Επομένω, είναι κάτι που θέλουμε εμεί από τη δική μα πλευρά να το ενθαρρύνουμε. Ευχαριστώ. Εμεί σα ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο, για τόσα μα εξηγήσετε. Οπότε ολοκληρώσαμε την ε, ακρόασή μα. Αλλά τώρα θα δώσουμε στην κυρία Γκαρδία Θάμπελ την σκητάλη, ούτως ώστε να διατυπώσουν τα συμπράσματά τους από όσα ακούσαμε και έτσι να ολοκληρώσουμε την τόσο ενδιαφέρουσα συνάντηση για να μάθουμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε το δρόμο για τους στόχους που αφορούν συγκεκριμένα τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ για δημιουργία απασχόλησης αλλά και ανάπτυξης. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Κατηθάμπαλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλου όσου έλαβαν τον λόγο. Ο στόχο τη ακρόαση ήταν να ακούσουμε όλους τους εμπλεκόμενους στην διαχείριση αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων, εργαλείων συγγνώμη, για την χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Δεν είναι θέμα συμπερασμάτων, αλλά ε, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι κάποια πράγματα αναδείχθηκαν επανειλημμένα κατά τη συζήτηση και πρόκειται για κάποιες έννοιες που και χθε ανέγυψαν. Μιλούσαμε για το χρηματοοικονομικό πλαίσιο ε, και μιλούσαμε για το σχέδιο ευρωπαϊκών ε, επενδύσεων, η προσθεμένη αξία, η απλούστευση ε, και αυτά λέγαμε χθε και η αλήθεια είναι ότι πέραν της απλούστευση έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά έχουμε επίσης την προσθεμένη αξία των χρηματοδοτικών εργαλείων που τώρα είναι ακόμα καλύτερη. Και επίσης έχουμε και όλα αυτά τα στοιχεία που δείχνουν ότι λειτουργεί το σύστημα αυτών των εργαλείων. Και αν συνεχίσουμε προς την απλούστευση, εάν συνεχίσουμε να περιχαρακώνουμε καλύτερα αυτά τα εργαλεία για να αποδίδουν περισσότερη ε, να πούμε περισσότερο, έχουμε και το θέμα το τρίτο που είναι η ευελιξία. Ε, και αυτή την ευελιξία την αποκτήσουμε να κάνουμε τα προηγούμενα. Τα ακούσαμε αυτά από το Ταμείο Επενδύσεων και από την Τράπεζα Επενδύσεων. Οπότε θα είναι καλύτερη η απόδοσή τους και άρα θα πρέπει να εργαστούμε σε αυτό το πλαίσιο για τα εργαλεία αυτά και έτσι και θα με αυτό το πνεύμα να κάνουμε την αναθεώρηση του πολιτικού ε, πλαισίου. Θα εξετάσουμε τις ε, λεπτομέρειες όμως που επόμενους μήνες. Σήμερα είδαμε ε, τις αδρές γραμμές, να δούμε πώς θα βρούμε κάποιες λύσεις, να δούμε πώς όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα μετασχηματίσουμε σε έναν κανονισμό, σε πολιτικές, ούτως ώστε αυτά τα εργαλεία να στοχεύσουν ε, όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα τους στόχους η κυρία Ρίαντα. Και εγώ να ευχαριστήσω την ε, κυρία Γκαρδία Θάμπελ που οργάνωσε αυτή την εκδήλωση, αλλά βέβαια και τον πρόεδρο μας, τον κύριο Αρτουή. Θέλω να σας πω ένα-δύο πραγματάκια, δηλαδή να ε, ξεκαθαρίσουμε κάτι το οποίο αναφέρει για την τράπεζα της ε, Ισλανδίας. Είναι κάτι το οποίο με Τσίγκλησε θα πρέπει να σας πω, όσον αφορά την δανειδοτική δυνατότητα προς τις μη Οι επιδόσεις είναι τραγικές και γι' αυτό και έτσι ήρθε η τράπεζα ενώπιον των δικαστηρίων σε σχέση με το σύστημα που είχαν. Επομένως το θέμα ε, δεν ήταν ότι δεν δανείζανε, ήταν ότι είχαν δημιουργική λογιστική. Παραποιούσαν τα νούμερα. Και γι' αυτό είπαμε ότι ε, θέλουμε να δούμε όχι πώς θα βοηθούν τις εμπορικές τράπεζες, πώς έχουν ένα σωρό χρήματα τα οποία ενισχύονται. Αλλά δεν θα κάνουμε για τις ΜΜΕ και επομένως όλοι συμφωνούμε σοβαρά την απλούστευση. Άρα έτσι μπορούμε να συμπλέψουμε και για την αναθεώρηση του πολιτού πλαισίου με όριζοντα το 2020. Αυτό σαν μήνυμα είναι ξεκάθαρο και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Έτσι ε, γίνεται η δουλειά όταν έχουμε τους εμπλεκόμενους να προχωρούν ακριβώς από τη βάση προς την κορυφή και όχι το ανάποδο. Είδαμε τι αποδίδει και τι δεν αποδίδει. Τα έμαθα. Και τώρα θα μελετήσω περισσότερο, θα πρέπει να εντείνουμε τον διάλογο, να κάθε χώρα να πει ό,τι καλύτερο έχει. Δεν θα σας καθέσω άλλο, θα είστε όλοι ε, κουρασμένοι, οπότε καλό σας βράδυ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε και εγώ να προσθέσω τις δικές μου ευχαριστίες στις δικές σας. Αλλά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ε, κυρία Νηριάντα και την κυρία Καρδιά Σάμπαλ. Πού στο να κάνουμε αυτή την ε, συνάντηση για τη χρηματοδότηση των μειοφιλών. Μιλούμε για απλούστευση και εμείς από τη θέση μας ως ευρωβουλευτές, μια που πρέπει να νομοθετούμε, να συμφωνούμε στις οδηγίες, θα, θα πρέπει με μετόλμη να νομοθετούμε, γιατί πολλές φορές αντιφάσκουμε. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε περισσότερη συνέπεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους τους ελεγοντολόγους και τους προσκεκλημένους μας. και θέλουμε να επαναλέγουμε το ότι πιστεύουμε στις ΜΜΕ.